So, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Οπότε καλό θα ήταν να καθίσετε παρακαλώ, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Παρακαλώ. Για την ημερήσια διάταξη. μπορεί να κρυθεί με μία τροποποίηση ο κύριος Πυρίνσκι παρακάλεσε το σημείο 11 να το ε, συζητήσουμε τελευταίο. Ελπίζω να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε σχεδόν όλες τις γλώσσες, αλλά φιλανδικά, μαλτέζικα, σλοβακικά, σλοβενικά, λετονικά και λιθωνικά. Αυτά δεν έχουμε. Ε, υπάρχουν μόνο, ε, υπάρχει μόνο δυνατότητα να τα μιλήσετε. Έχουμε μία ομάδα επισκεπτών από την κυρία Αλεσάνδρα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια άλλη ομάδα επισκεπτών. Σήμερα στις ανακοινώσεις του Προέδρου προβλέπετε να σας ενημερώσω σύντομα για τις τρεις αντιπροσωπείες, τρεις αποστολές που είχαμε πρόσφατα. Πρώτα μία αποστολή στην Ολλανδία για την επερχόμενη Προεδρία Δεύτερον, προς τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας στη Γενέβη και τρίτη αντιπροσωπεία πήγε στην Πορτογαλία. Πολλά ταξίδια λοιπόν. Όλη αυτή η ιστορία έληξε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε τώρα πρέπει να σας ανακοινώσουμε τι έγινε. Αλλά προτείνω να μην γίνει σήμερα αυτό, για να μην ε, χάσουμε χρόνο και να ακούσουμε αμέσως ε, την κυρία Τάισεν, ε, την οποία χαιρετίζω και την ευχαριστώ που είναι στη διάθεσή μας για μια μισή ώρα. Αν συμφωνείτε λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτές τις αποστολές ε, στις 27 Ενδεκάτου ή 3 Δωδεκάτου. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Ωραία. Οπότε το μόνο θέμα που μένει είναι τα πρακτικά για 12 και 13 Οκτωβρίου. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία. Οπότε περνάμε ήδη στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Είναι παρούσα εδώ η κυρία Τάισεν για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής του 16 όπου υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν πολύ την Επιτροπή Απασχόλησης αλλά και κάποιες ανακοινώσεις ε, και ορισμένα τα οποία μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι προκύπτουν από τις ομιλίες του κυρίου Γιούνκερ, της κυρίας Τίσεν και όλα αυτά μας κάνουν να θεωρούμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε του χρόνου πολλά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν πολλή εργασία. Για παράδειγμα, ελάχιστες προδιαγραφές προσαρμογή προς τα πάνω, κινητικότητα των εργαζομένων στο αρχικό στάδιο και διάφορα άλλα θέματα για τα οποία θα θέλαμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων τόσο ώστε η Επιτροπή μας να μπορέσει να προετοιμαστεί σωστά για αυτά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ούτω ώστε σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαμορφώσουμε σωστά τα θέματα. Χωρίς λοιπόν να ε, μακρηγορήσω περαιτέρω να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τάισεν. Ελπίζουμε να ε, μιλήσετε 15 λεπτά, παρακαλώ, για να μην με, ε, μου γκρινιάζουν μετά τα μέλη της Επιτροπής μου ότι δεν τους άφησα χρόνο να μιλήσουν και εκείνοι. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Αξιότιμα μέλη. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που είμαι μεταξύ σας. Είναι ένας χρόνος από τότε που ανέλαβε η νέα Επιτροπή. Τον Οκτώβριο του 2014, κατά την ακρόασή μου, ενώπιόν σας, ε, παρουσίασα τους στόχους μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και επενδύσεις σε καλύτερη κοινωνική προστασία. Δηλαδή να επενδύσουμε σε καλύτερη κοινωνική προστασία. Παρά τα πολλά χρόνια, τα πέντε χρόνια βαθιάς οικονομικής κλίσης, κρίση, συγγνώμη, τώρα βλέπουμε κάποια, κάποια μηνύματα θετικών εξελίξεων. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2014, ο αριθμός των ανέργων έπεσε κατά 1,5 εκατομμύριο ατόμων στην Ευρώπη των 28 και, τα, και κατά 900.000 άτομα στην Ευρωζώνη. Όμως δεν είναι ομοιόμορφη αυτή η πτώση της ανεργίας. Έχουμε ανεργία 9,5% στην Ευρώπη των 28, αλλά βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις από 4,5% μέχρι 25% η χαμηλότερη ανεργία. Τον ε, παρελθόντα Αύγουστο ήταν στη Γερμανία 4,5%, Τσεχία 5%, Μάλτα 5,1% και η υψηλότερη ανεργία ήταν 25,2% στην Ελλάδα και 22%, 22 στην Ισπανία. Αλλά η μείωση της ανεργίας σημειώνεται σε 23 κράτη-μέλη. Αυτοί που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό επίσης μειώθηκαν σταδιακά από 124 εκατομμύρια το 2012 σε 121,8 το 2014. αλλά δεν επιτύχαμε το στόχο μας γιατί στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Ε, Επανέρχεται λοιπόν ε, η ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν. Η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί και θίγει 12 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 60% είναι άνεργοι για δύο χρόνια ή παραπάνω. Και, και πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετωνία, Λιθουανία και Ουγγαρία απειλεί το το 2013 από κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτό το ποσοστό ήταν 15-16% στη Σουηδία, την ε, Ολλανδία και την Τσεχία. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε αποκλήσεις. Αυτές οι αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών συνοδεύονται και από αποκλήσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών. Και αυτό είναι μεγάλος λόγος ανησυχίας γιατί απειλούν την συνοχή των κοινωνιών μας, την ανταγωνιστικότητά μας και τη δυνατότητα ανάπτυξης της Ευρώπης. Στο πρώτο έτος της νέας Επιτροπής εργαστήκαμε σκληρά για να ε, επιτύχουμε τους στόχους ε, εφαρμόζοντας ε, το πρόγραμμα εγγύσεων για την εργασία των νέων και αυξήθηκε η προχρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό, ούτω ώστε επιτόπου τα προγράμματα να αρχίσουν να λειτουργούν πιο σύντομα. Και επίσης υπήρξε και σύσταση για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Και τρίτον, έχει υπάρξει μια νέα στον πανευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην ανάπτυξη Τη ε, κοινωνική πολιτική και τη πολιτική απασχόληση και δεσμεύομαι πλήρω να υπάρξει περαιτέρω αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Αλλά σαφώ. δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα πράγματα έχουν επανέλθει σε ομαλή κατάσταση και το επόμενο δωδεκάμινο η δράση μα θα καθοριστεί από αυτό το πλαίσιο. Να εστιάσω σε μερικού άξονε όπου θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά για να επιτύχουμε αποτελέσματα και προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία. Πρώτον, Έχουμε τον πυλώνα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της οικονομίας της αγοράς μας. Είναι μία από τις κύριες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Η κρίση έχει αφήσει ε, τις σουλές και πολλοί είναι σε επισφαλή απασχόληση, ε, αγωνίζονται να βρουν εργασία. Και ο κόσμος της εργασίας επίσης το περιβάλλον της εργασίας αλλάζει ταχύτατα, αυτό σημαίνει νέες ευκαιρίες αλλά και νέα ερωτηματικά. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστώ για ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το κοινοτικό κεκτημένο θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και θα παραμείνει ισχυρό στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Θέλουμε η νομοθεσία μας να συντονίζεται με τις ε, πραγματικότητες της σύγχρονης ζωής, ο συνδυασμός της εργασίας και της οικογενειακής, εργασίας, και της οικογενειακής ζωής, ε, η τηλεργασία κτλ. χωρίς να παρεμποδίζεται η ε, ελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Πρέπει να δώσουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά πρέπει επίσης να στηρίξουμε τους εργαζόμενους για να προσαρμοστούν και να τους παράσχουμε επαρκή προστασία όταν τη χρειάζονται. Ο στόχος μας είναι να μειωθεί η επισφαλής εργασία, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης για θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Οι αυξανόμενες αποκλήσεις μεταξύ κρατών μελών είναι τεράστιος λόγος ανησυχίας. Υπονομεύει μία από τις βασικές αιτίες ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την κοινωνική σύγκληση και τη βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαίων. Γι' αυτό ο κύριος στόχος μας πρέπει να είναι η κοινωνική σύγκληση προς τα πάνω. Ο στόχος μας είναι να έχουμε προδιαγραφές ευρέως συμφωνημένες για την εργασία που να ενισχύσουν τη σύγκληση παντού στην Ευρώπη. Πρέπει αυτά οι προδιαγραφές ε, να εφαρμόζονται και σε καλούς και σε κακούς καιρούς. Αυτές οι τιμέ αναφορά θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές μας για να ενθαρρύνουμε μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη με βάση την εγγύηση για την νεότητα και την ε, καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας στα πλαίσια ακριβώς της ενίσχυσης της ΟΝΕ γιατί όπως ξέρετε στα πλαίσια της ΟΝΕ υπάρχει υψηλότερη αλληλεξάρτηση των κρατών μελών για την αμοιβαία ευημερία. Θα υπάρξει λοιπόν ενισχυμένο διάλογος προς την κατεύθυνση αυτή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους. Για να υπάρξει αποτελεσματική μεταρρύθμιση της πολιτικής. Και θα οργανώσουμε αυτό το διάλογο ούτω ώστε να υπάρχουν συντονισμένες προσπαθίε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι αναγκαίο. Δεύτερο, πολύ σημαντικό για την επόμενη χρονιά, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την απασχόληση, την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας. Εξετάζουμε το κεκτημένο στον τομέα αυτό, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε μια απλουστευμένη αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στόχος μας είναι να υπάρχει μια απλουστευμένη δομή που να καθορίζει σαφέστερα το κεκτημένο, να μειώσουμε τον αριθμό των οδηγιών ενώ παράλληλα θα διατηρήσουμε το επίπεδο προστασία σε υψηλό επίπεδο και πρέπει να ενισχύσουμε επίση την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων περαιτέρω με βάση τι πρόσφατες επιστημονικέ εξελίξει. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν πεθαίνουν εργαζόμενοι, όταν κατασκευάζουν τα καταναλωτικά μας αγαθά ή όταν ε, υφίστανται νέους κινδύνους, εκτίθενται σε νέες καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες. Έτσι λοιπόν, πριν το επόμενο καλοκαίρι θα προσθέσουμε, θα προσθέσουμε περισσότερες ουσίες στον κατάλογο των ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, τις καρκινογενείς ουσίες και τις ε, ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις. Θέλουμε όμως παράλληλα να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια αγορά με ταχεία τεχνολογική εξέλιξη και ταχαίως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Γι' αυτό οι επιχειρήσεις μας πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καινοτομίε, να επεκταθούν και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τις σωστές δεξιότητες για να ανταποκριθούν στην αλλαγή στην ζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν εργαζόμαστε για ένα θεματολόγιο δεξιοτήτων για να βελτιώσουμε την απασχολησιμότητα των εργαζομένων μας, να διασφαλίσουμε την αναγνώριση και δυνατότητα μεταφορά από χώρα σε χώρα των δεξιοτήτων του και των πτυχίων τους και να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ εκπαίδευση και κόσμου τη εργασία και των επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι οι δεξιότητε που χρειάζονται τώρα οι εργαζόμενοι είναι πολύπλοκε και συνδυασμένε, Για παράδειγμα, ε, πληροφορική ε, χρήση μηχανημάτων. Και ξέρουμε επίση ότι η οικονομική κρίση έχει καταστρέψει πολλέ θέσει εργασία, ιδιαίτερα των ε, εργαζομένων χαμηλών δεξιοτήτων, ενώ οι περισσότερε νέε θέσει εργασία χρειάζονται διαφορετικέ δεξιότητε και πιο περίπλοκες, υψηλότερο επίπεδου. Οι ψηφιακές δεξιότητες ε, γίνονται όλο και πιο αναγκαίες στην οικονομία μας και σίγουρα θα είναι προτεραιότητα. Αλλά για να βοηθήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητε, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν ένα βασικό επίπεδο δυνατότητας χρήσης της γλώσσας και μαθηματικών δεξιοτήτων. Πολλοί Ευρωπαίοι έχουν μόνο χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων σε αυτούς τους δύο τομείς. Και ένας στους 15 νέους δεν τα πάει καλά σε πολύ βασικές δεξιότητες. 40% των πολιτών μας έχουν μόνο πολύ χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές δεξιότητες. Πρέπει να αυξηθούν λοιπόν αυτές τις δεξιότητες όχι μόνο για την εργασία, αλλά και για τη ζωή του κάθε ατόμου είναι όντως η οδός προς την ευημερία γιατί δίνει και δυνατότητες απασχόλησης και δυνατότητες ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Είναι προφανές ότι πρόγραμμα για να βοηθήσουμε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα βοηθούν τους νέους και ευνοούν τη δυνατότητα εξέβρεση εργασίας. Πρέπει λοιπόν η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να είναι πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή. Καταλήγοντας από αυτού πρέπει να επενδύσουμε στους εργαζόμενούς μας. Η ανταγωνιστικότητά μας βασίζεται κυρίως στον επιτυχή συνδυασμό καινοτόμων επιχειρήσεων και υψηλά εκπαιδευμένων και παραγωγικών εργαζομένων. Και τώρα να στραφώ προς τη νέα αρχή για τους εργαζόμενους γονείς. Αυτή η νέα πρωτοβουλία χρησιμοποιεί την ε, πρόσφατη απόσυρση της ε, πρότασης ε, για την άδεια μητρότητας και δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπιση σε ευρύτερο πλαίσιο τα διάφορα προβλήματα που έχουν, να, που έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η νέα προσέγγιση θα είναι υποφελής για όλους, ειδικότερα για τις γυναίκες ε, την συμμετοχή του στην αγορά εργασίας. Ε, ε, επίσης θα μειωθεί το χάσμα στις συντάξεις και γενικότερα θα είναι καλύτερο για την κοινωνία αλλά και για τους υπεύθυνους φροντίδας οι οποίοι είναι επίσης πολύ σημαντικοί στην κοινωνία και τα παιδιά θα ε, διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο να ζήσουν στη φτώχεια. Όπω ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλέ φορέ τονίσει τη σημασία τη ύπαρξη πολιτικών και για του πατέρε εκτός από τι μητέρε, η νέα πρωτοβουλία θα εξετάσει πώ μπορούμε ισότιμα να χρησιμοποιηθεί ε, ένα καλύτερο διακανονισμό γονεϊκή άδεια. Οι ανάγκε των ανθρώπων που έχουν εξαρτώμενα μέλη μεγάλη ηλικία. Ε, ή απλώς εξαρτώμενα μέλη, ε, επίσης θα ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα να αναφερθώ κύριε Πρόεδρε στα ε, όσα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Εμείς αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε την προπαρασκευαστική μας εργασία για την κινητικότητα της εργασίας ε, για την οποία θα παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία μας τον επόμενο μήνα. 2 Δεκεμβρίου θα γίνει η έγκριση, πριν, μία μέρα πριν ε, από την ε, Διεθνή, την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες. Μετά το θέμα των μακροχρόνια άνεργων, μια ανακοίνωση η οποία, μια ανακοίνωση η οποία θα εγκριθεί στις 12 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ και ελπίζουμε κατά τις επόμενες εβδομάδες να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, το Eures και την πλατφόρμα κατά της αδήλωτης εργασίας, κάτι το οποίο απασχολεί και εσάς. Έχει πλέον υπάρξει συνένεση στον τριμερή διάλογο και ελπίζουμε ότι εντός του τρέχοντος έτους θα υπάρξει συμβιβασμός. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, δεν είναι ομαλή η κατάσταση των πραγμάτων, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το κοινωνικό αντίκτυπο της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και τα, ε, με τα διαρθρωτικά προβλήματα της ε, γυράσκουσας, ε, του γυράσκοντος εργατικού δυναμικού μας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ενσωμάτωσης χιλιάδων ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία. Επομένως, ε, Νέες προκλήσεις ε, απαιτούν νέες ευρωπαϊκές ε, συντονισμένες λύσεις είναι δική μας ευθύνη να ε, λύσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα για να ε, μπορέσουμε να επιτύχουμε την κοινωνική ένταξη, κάτι το οποίο θα μπορέσει να δώσει στην κοινωνική Ευρώπη τη νέα αρχή που χρειάζεται. Χρειάζεται επίσης ε, να υπηρετήσουμε όλους τους πολίτες μας με αποτελέσματα, δίνοντάς τους πραγματικές ευκαιρίες και προστασία. Δεν μπορούμε να χτίσουμε την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζούμε αν ε, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιες αγορές ε, και αν δεν έχουμε ισχυρή κοινωνική συνοχή. Πρέπει να ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη όπως επίσης και την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αυτή είναι η δική μου θεώρηση προκειμένου κοινωνικά η Ευρώπη να είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και με πολύ χαρά θα απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ θερμά για το πρώτο μέρος της συζήτησής μας και αυτά που μας είπατε. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα ακούσουμε τους συντονιστές. Ο καθένας θα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Και κατόπιν θα ζητήσουμε από την κυρία Τάισεν να απαντάει σε ένα λεπτό κάθε φορά πριν πάρει το λόγο ο επόμενος. Αυτή η διαδικασία ζητήθηκε και γι' αυτό δίνω το λόγο καταρχάς στον David Κάζα. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Καλημέρα σε όλους. Η Επιτροπή πώς σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία με εθνικούς και περιφερειακούς φορείς για να φτάσει στους πολίτες που χρειάζονται πόρους για να βελτιώσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι απλά να δημιουργούμε νέους πυλώνες. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής και αποτελεσματικής απορρόφησης των πόρων, ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές περιοχές. Ευχαριστώ. Εντυπωσιάστηκα. Ja, danke schön. Η κυρία Τάισεν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι περισσότεροι από τους πόρους μας είναι αντικείμενο κοινή διαχείρισης. Πρέπει να συνεργαζόμαστε λοιπόν με τα κράτη-μέλη. Τα κρατη μελη συμβάλλουν σημαντικά στην ε, εκτέλεση των προγραμμάτων. Καταρχάς φροντίζουμε τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί να ταιριάζουν στο νομοθετικό πλαίσιο και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Και παρακολουθούμε από κοντά το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά, το πώς δαπανώνται. Και δεν ελέγχουμε απλά αν έχουν δαπανηθεί για τον στόχο τους, όπως κάναμε πριν μερικά χρόνια. Όπως γνωρίζετε, έχουμε τώρα μία νέα προσέγγιση στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενισχύουμε αυτήν τη νέα προσέγγιση μας. Δεν εξετάζουμε δηλαδή μόνο αν έχουν δαπανηθεί οι πόροι σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά ε, βλέπουμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θέλουμε να ακούσουμε τις περιφέρειες, τα κράτη-μέλη που δαπανούν τα χρήματα αυτά, ε, για να μας πούνε ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Γιούτα Στάινρουκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τις ε, παρατηρήσεις σας. Η Κομισιόν χρειάστηκε αρκετό χρόνο για την ε, προετοιμασία της νομοθεσίας. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τα κοινωνικά δικαιώματα. Μιλήσατε για περισσότερη ευελιξία των εργαζομένων. Θα είναι απαραίτητη όμως και περισσότερη προστασία. Ποιοι είναι συγκεκριμένα οι στόχοι σας. Θέλετε να ενισχύσετε την σύγκληση. Ποια είναι τα συγκεκριμένα σας μέτρα στο θέμα αυτό. Ο κύριος Γιούνκερ αναφέρθηκε στην αρχή ε, ίση αμοιβή για, για την ίδια δουλειά στον ίδιο τόπο. Και το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα του για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν ζήτησε ο όρος του εργαζόμενου να οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν νέες μορφές απασχόλησης ε, λόγω της ψηφιοποίησης, ε, για παράδειγμα, στην Γερμανία. Έχουμε όλο και περισσότερου ε, ανεξάρτητους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό εξαρτάται από ε, τους κρατικούς πόρους που διατίθενται σε κάποιους τομείς. Η Κομισιόν πώς το βλέπει αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τάισεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εντός ενός λεπτού. Όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, έχουμε εδώ δύο σκέλη υπάρχουν κάποια βασικά κοινωνικά δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη μπορούν να πάνε πιο πέρα. Πρέπει όμως να εγγυώνται κάποια ελάχιστα δικαιώματα και θα πρέπει να εξετάσουμε εάν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία στην εργασιακή ζωή και αν υπάρχουν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουμε σχετικές προτάσεις. Μιλήσατε επίσης για τον ορισμό του εργαζόμενου. Μπορεί να μην έχουμε υποβάλει ακόμα πρόταση, το εξετάζουμε όμως. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εταιρείας Uber. Τι ακριβώς είναι ο εργαζόμενος, τι προστασία πρέπει να έχει. είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα επανεξετάσουμε. Όσον αφορά την σύγκληση, δεν έχουμε εντολή στο θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη θέλουν όμως να συγκλίνουν μεταξύ τους σε κάτι το οποίο έχει αρνητικέ συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν με τα κράτη-μέλη, με τους κοινωνικού εταίρους να συμφωνήσουμε καταρχάς όσον αφορά τους στόχου και σε δεύτερη φάση να υποβάλουμε συστάσεις, ε, κάτι που άλλωστε κάναμε και για την εγγύηση για την νεολαία. Με την διάθεση πόρων θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την ανάπτυξη και να εργαστούμε με στόχο την μεγαλύτερη σύγκληση. Όσον αφορά την ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά, ο κύριος Γιούνκερ το ανέφερε αυτό επανειλημμένα και χαίρομαι γι' αυτό, διότι συμφωνώ απολύτως. Είναι μια ιδέα που αναφέρεται κυρίως στην απόσπαση εργαζομένων. Έχουμε τη σχετική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τις περιπτώσεις σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην αμοιβή ανδρών και γυναικών. Αυτό πάντως ε, έχει να κάνει με το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι τελείωσε το λεπτό που είχα στη διάθεσή μου. Δεν ξέρω αν υπήρχε και άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Ε, η κυρία Στάινρουκ, ε, δεν εξέλιξα το χρόνο μου. Μία τελευταία ερώτηση λοιπόν εμφανίζονται όλο και περισσότερες νέες μορφές εργασίας, για παράδειγμα με την ψηφιοποίηση. Έχουμε όλο και περισσότερους ε, ελεύθερους ανεξάρτητους επαγγελματίε, ε, που ε, χρειάζονται όμως χρηματική βοήθεια. Μήπως θα μπορούσατε να απαντήσετε στο θέμα αυτό. Η Επίτροπος, θα απαντήσω πολύ σύντομα είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με τον ορισμό του εργαζομένου. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις προϋποθέσεις το πώς αλλάζουν οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες εργασίας και θα πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα τον ορισμό. Διότι είναι πια απεπαλαιωμένος ο ορισμός σε κάποιους τομείς. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τις νέες εξελίξεις, να εξετάσουμε τι είναι ο εργαζόμενος, ε, τι είναι ο ελεύθερο επαγγελματίας, διότι υπάρχουν ε, άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίε ε, που εξαρτώνται από έναν μόνο εργοδότη. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις νέες εξελίξεις και θα δούμε αν μπορούμε να υποβάλουμε σχετικές συστάσεις. Ευχαριστώ Τόνας. Όχι. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν Αντέα δεν είναι σωστός ο καταλογός μου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Καταρχάς, χαιρετίζω αυτή την προσέγγιση που έχετε καλύτερων ρυθμιστικών μέτρων. Σημαντικό λοιπόν να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και το συνδέω αυτό με αυτά που είπατε για την απλούστευση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια διασφαλίζοντας ότι διατηρείται το επίπεδο προστασίας που θέλουμε αλλά μέσω απλωστευμένων διαδικασιών ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες να τηρούν τους κανόνες. Η ερώτησή μου αφορά κάτι που δεν αναφέρατε. Δηλαδή, η αναθεώρηση, η επανεξέταση τις οδηγίες για τις αποσπάσεις. Ακούσαμε πολλά για αυτό το θέμα. Θα με ενδιαφέρε ιδιαίτερα να μάθω εάν σε αυτή τη φάση θα υποβάλλεται ή όχι κάτι. Γιατί ελπίζω να μην υποβάλλεται νέες προτάσεις, γιατί θεωρώ ότι σε αυτή τη συγκυρία το σημαντικό είναι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η οδηγία για την εφαρμογή της οδηγίας για την ε, απόσπαση. Εάν λοιπόν ξανοίξουμε το θέμα της αρχικής οδηγίας πριν εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία εφαρμογής, τότε θα δαπανίσουμε πολύ κόπο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις χωρίς να δούμε πώς ακριβώς εφαρμόζεται το αρχικό κείμενο. Νομίζω πως θα ήταν σοβαρό λάθος να επανέλθουμε επί της αρχικής οδηγίας. Και σε σχέση με αυτό, ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας. Βεβαίως είναι ευγενέστατος στόχος. Και στη χώρα μου έχουμε ένα νόμο για το θέμα των αμοιβών αναφύλων. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η καλύτερη κανονιστική προσέγγιση είναι δύσκολη σε αυτό τον τομέα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 250.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στα Βρετανικά δικαστήρια για το θέμα αυτό. Πώς εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία για την ίση αμοιβή στον ίδιο τόπο και ανησυχώ πολύ για την οδηγία για τους ε, αποσπασμένους γιατί στον τομέα των υπηρεσιών αν αποσπάσεις κάποιον για παράδειγμα από τη χώρα μου στην Ουγγαρία για παράδειγμα όπως ε, έχω κάνει εγώ η ίδια αν πεις ότι πρέπει να πληρωθούν το ίδιο ή θα πρέπει να τους πληρώσω με ουγγρικούς μισθούς και δεν θα πάνε τότε ή παρεβαίνουμε στις εθνικές διαπραγματεύσεις για τις αμοιβέ, κάτι το οποίο θα ανησυχήσει πολύ τον κύριο Όρμπαν. Ενδιαφέρον ερώτηση, λέει πρόεδρος αλλά μακρηγορήσατε κάπως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Μακιντάιρ λέει η κυρία Τάισον. Η απλούστευση. Η προσπάθειά μας ε, συνεχίζει, έχουμε ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Γιατί είμαστε πεισμένοι ότι είναι αναγκαίο. Θα το κάνουμε όπως ήδη ανέφερα. Θα προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε, απλουστεύσουμε την πληροφόρηση που δίνουν οι μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις για στατιστικούς λόγους. Γιατί και εδώ είναι ε, πολλά αυτά που πρέπει να κάνουν. Και θέλουμε να απλωστευθεί και η διαδικασία λογοδοσίας για τις χρηματοδοτήσεις που δίδονται από τις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες, τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να διευρυνθεί η δυνατότητα της απλουστευμένης ε, επιλογής για την αποτίμηση και λογοδοσία για το κόστος, για την απόσπαση των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας. Έχετε δίκιο. Η μεταγραφή της οδηγίας εφαρμογής είναι πολύ σημαντική και η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε πολλά προβλήματα με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και γι' αυτό εγκρίναμε αυτή τη νέα οδηγία εφαρμογή, ούτω ώστε να έχουμε τώρα δύο οδηγίες. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. πριν τα μέσα του 16 γιατί αυτό είναι το όριο και τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν με ποιοτικό τρόπο αλλά υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμη επιληθεί και δεν θα επιληθούν και μέσω της ε, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο αυτής της οδηγίας, εφαρμογής της απόσπασης. Γι' αυτό εξετάζουμε και την ίδια την οδηγία απόσπασης για να δούμε μήπως μπορούμε να βελτιώσουμε, μήπως πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα θέματα με στόχο συγκεκριμένα. Να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι πολίτες σε κάποιες χώρες δεν θεωρούν ότι αντιμετωπίζονται δίκαια οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι και το διαπιστώνουμε και εμείς αυτό. Και γι' αυτό και με πολλή στήριξη από τον πρόεδρο της Επιτροπής επανήλθαμε σε αυτή τη βασική έννοια η ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας. Ξέρω, αυτό δημιουργεί δυσχέρειες. Και πολλοί προσφεύγουν στα δικαστήρια για να διευκρινιστεί η νομική κατάσταση. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο που δεν θα είναι ε, επανεπινόηση του τροχού. Προσπαθούμε να δούμε τι υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, υπάρχει νομολογία εκεί. Άρα, πώς να το πω, να διευκρινίσουμε τα νομικά θέματα, αν υπάρχει νομική ασφάλεια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό ήθελα να πω. και για τους εθνικούς μισθούς, τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των αμοιβών. Όχι, δεν παρεμβαίνουμε σε αυτό. Το μόνο που ζητάμε είναι αν κάποιος εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος, όπου αναφέρεται στην νομοθεσία ότι η ελάχιστη αμοιβή πρέπει να γίνεται σεβαστή, να γίνεται. Αλλά δεν θα παρέμβουμε στον καθορισμό των αμοιβών στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και σε πολλά κράτη-μέλη αυτό έχει εκχωρηθεί στους κοινωνικούς εταίρους και αυτό θα το σεβαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ούλα Τόνετς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν την αναθεώρηση της οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων γιατί ακόμα παραμένει ασαφές για μένα τι είδους ε, αναθεώρηση θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν δούμε ε, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρει ακριβώς αυτό που είπε μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ίδια πρέπει η ίδια αμοιβή ε, και για τα δύο φύλλα σε ίδιο τόπο. Οπότε αυτή, αυτή η αναθεώρηση σε αυτό πρέπει να προσβλέπει. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει λίγο περισσότερα σε σχέση με τις ιδέες που εξεργάζεται αυτή τη στιγμή ε, για το θέμα της απόσπασης εργαζομένων και το θέμα του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα και επ' αυτού πώς θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της νομικής βάσης στις διάφορες ε, συνθήκες στις οποίες βασίζεται ε, αυτό. Έχετε το λόγο. Αγαπητή συντονίστρια, φαντάζομαι ότι σας απασχολεί πάρα πολύ το περιεχόμενο των προτάσεων ε, σε σχέση με την απόσπαση και τον συντονισμό των, κοινωνικών ασφαλίσεων, των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων. Ε, το συζητούμε ε, αυτό εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε μία συζήτηση προς ανατολισμού την οποία έχουμε ήδη κάνει. Εγώ υποστήριξα τους συναδέλφους σε σχέση με αυτό το θέμα της ίσης αμοιβή, οπότε πρέπει να επιστρέψω στο σώμα των επιτρόπων και να δω κατά πόσο υπάρχει συμφωνία επ' αυτού. Είμαι πάντως βέβαιη ότι θα βρούμε μία σωστή λύση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε πολλούς τομείς είναι κάτι το, με το οποίο έχουμε συνηθίσει να εργαζόμαστε στο πλαίσιο της νομοθεσίας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο επίσης ε, θα εξετάσουμε όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων και την απόσπαση είναι το εξής. Πρέπει να δούμε την έννοια της προσωρινής εργασίας, της προσωρινής διάρκειας της απόσπασης. Γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, δεν υπάρχει συνοχή ε, με την κοινωνική ασφάλιση, το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης παρακολουθούμε πολύ στενά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και στο πλαίσιο της ε, ε, παροχής ασφάλειας δικαίου. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό όσον αφορά τον πυλώνα των κοινωνικών δικαίων Πώ Πώς θα οργανώσουμε το να ληφθεί υπόψη η νομική βάση ε, της συνθήκης. Δεν θέλουμε να υπερβούμε τις αρμοδιότητές μας. Εμείς ε, σεβόμαστε τους κανόνες, σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας και θα υποβάλουμε προτάσεις μόνο ε, στους τομείς στους οποίους έχουμε αρμοδιότητα. Υπάρχουν όμως κάποια ζητήματα για τα οποία μπορούμε να υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις γιατί έχουμε αρμοδιότητα ε, βάσει του άρθρου 153 της συνθήκης. Ε, για άλλους τομείς χρειαζόμαστε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και το συντονισμό των πολιτικών και είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε για τη συγκριτική αξιολόγηση. Εκεί θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία μέθοδο ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε συγκεκριμένους στόχους και να οδηγήσουμε τους εταίρους στο να ε, επιτύχουν αυτούς τους στόχους, να αποδεχθούν την ε, ε, αναθεώρηση των ομοτήμων, όπως επίσης και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης. Βεβαίως θα σεβαστούμε την νομική βάση και τις συνθήκες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κούνεβα τώρα για την ΚΟΥΑ. Α, δεν θα μας μιλήσει η κυρία Κούνεβα. Ωραία, θα αντιστρέψουμε τη σειρά. Η πράσινη λοιπόν. Η συνάδελφος Στάνοκα. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε σε ένα πακέτο κινητικότητας εργαζομένων για την μείωση της ανεργίας. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα είναι όταν πηγαίνει κάποιος από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και εγώ προέρχομαι από τη Λετωνία όπου πολλοί κόσμος το κάνει αυτό. Τα κοινωνικά δικαιώματα μειώνονται, υπάρχουν διακρίσεις και ε, υπάρχουν κοινωνικές αντικσοότητες είναι άσχημο να κατηγορούμε ε, τους πολίτες επειδή απλώς ασκούν ε, τα θεμελιώδη ε, δικαιώματά τους αναζητώντας εργασία κάπου αλλού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε και να προστατεύσουμε αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα εργασίας κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αντιμετωπίσετε τη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, όσον αφορά την περιορισμένη πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τίσεν. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ο, ποιος είναι ο στόχος ε, του πακέτου κινητικότητας και των πρωτοβουλειών ε, που θα υπάρξουν στο πλαίσιο αυτό. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε τη διευκόλυνση και την ε, ε, ενθάρρυνση της κινητικότητας, η οποία είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι ένας πυλώνας της εσωτερικής αγοράς μας, ε, μας οδηγεί στην ανάπτυξη, δίνει ευκαιρίες στον κόσμο, δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να βρουν θέσεις εργασίας και στις δικές τους χώρες και επίσης γίνεται αντιστοιχεία αναγκών και δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε συνεχίσουμε να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας ε, όταν μιλούμε για την κινητικότητα των εργαζομένων, πρέπει να <clears throat> εξασφαλίσουμε ότι όσοι ασκούν το δικαίωμα της κινητικότητας ε, να μπορούν να χαίρουν της απαραίτητης <coughs> προστασίας ε, στο πλαίσιο των διαφόρων θεσμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρηθεί όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας. Αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι πολίτες ε, να ε, συμμετέχουν στα προγράμματα ανεργίας και στη χώρα τους να εξασφαλίζεται ότι ε, μπορούν να μεταφερθούν τα δικαιώματά τους. Αν κάποιος πάει σε μία άλλη χώρα για να αναζητήσει εργασία, να μην βρεθεί σε ένα κενό εντός του οποίου δεν θα μπορεί να έχει δικαιώματα ούτε βάσει του ενός ούτε βάσει του άλλου συστήματος. Επομένως πρέπει ε, να δούμε κατά πόσο τα επιδόματα της χώρας προέλευσης μπορούν να διατηρηθούν στη χώρα υποδοχής. Αυτό είναι, γι' αυτό είναι σημαντικό ο συντονισμός, να μην υπάρχουν μαύρες τρύπες. Πρέπει κάθε φορά ε, οι πολίτες να μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους και να είναι επιλέξιμοι στο ένα ή στο άλλο κράτος. Ελπίζω αυτό να καλύπτει το ερώτημά σας. Και τώρα η Κωνσταντίν Κακούνευα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κυρία Επίτροπε, στην ομιλία σας εδώ μας είπατε πράγματα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα της Επιτροπής το 2016. Αποτιμώντας λοιπόν συνολικά το πρόγραμμα, θα ήθελα να ρωτήσω. Είναι δυνατόν όταν η Επιτροπή απαριθμεί την ανάληψη διαφορετικών δράσεων για το όραμά σας η εργασία να κατάσετε τελευταία και πάλι πίσω από τα οικονομικά θέματα και θα σας προλάβω. Ξέρω πολύ καλά πως η Επιτροπή είναι και μια αγορά. Η Επιτροπή όμως είναι και οι πολίτες της. Και τα τελευταία χρόνια η οικονομία έχει πνίξει τους πολίτες της γιατί δεν αναπτύσσεται προς όφελος τους. Αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας τους ως μέσα και όχι ως αποδέκτες του πλούτου της. Μη μου πείτε πως η ανάπτυξη άλλων πολιτικών θα βοηθήσει της απασχόληση γιατί να δεν υπάρχει έστω και φράση που όμως είναι θεμέλιο των συνθηκών για κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Οι πολίτες θα αποφυληθούν από την πολιτική για την ε, κινητικότητα όπως αναφέρεται και από μια αναθεωρημένη οδηγία που ακόμα δεν έχουμε δει για τις αποστάσεις των για τις αποσπάσεις των εργαζομένων και αν ετοιμάζεστε να μου πείτε πώς η ανάπτυξη άλλων τομέων τα φέρει εργασία θέλω να μας περιγράψετε γιατί τι είδους εργασία μιλάμε. Στην Ελλάδα ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του και να μην παίρνει στις συντάξεις να μας δίνετε έκτακτης χρήματα για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης αλλά σε ποιο πλαίσιο φαντάζομαι πως έχετε διαβάσει την έκθεση που δημιουργήσε η ίδια επιτροπή της Ευρώπης στις αρχές του χρόνου για τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη. Ε, εκεί σημειώνεται πως σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από την κρίση οι εργασιακές σχέσεις άλλαξαν με διαφορετικούς τρόπους εντονότερα, ταχύτερα και συχνότερα. Πώς δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιες μεταβολές είναι προσωρινές και ποιες είναι πιθανώς μόνιμες. Πώς η μορφή που τα πάρει ο κοινωνικός διάλογος μετά την κρίση εκκρεμεί ακόμα αποτυπώσει αντίκτυπος της κρίσης και η δημοσιονομική εξυγίανση που εφαρμόστηκε σε πολλές χώρες άσκησε πιέσει στον κοινωνικό διάλογο με διάφορους τρόπους. Τα επισυνά το απίστευτο είναι πως η Επιτροπή με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχω αναπήρει και δεν μπορώ να μιλήσω πιο γρήγορα λέξει και οι σελίδε είναι όσο η τελευταία κανονική ομιλία. Νομίζω ότι έχω δικαίωμα να μιλήσω ακόμα λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το απίστευτο είναι πω η Επιτροπή παραδέχεται πώ η επίγουσα ανάγκη πρόθεση αυτών των ταχαίων αλλαγών επιβλέπει στην τόνιση της οικονομικής μεγέθυνσης. Η Επιτροπή παραδέχεται επιπλέον πως η φιλοσοφία αυτή, η αποδυνάμωση των συνολικών συμβάσεων εξυπηρετεί την ευθυγράμμιση μισθών και παραγωγικότητας και πως οι αλλαγές στα συστήματα κατορισμού των μισθών στα κράτη-μέλη που ακολουθούν πρόγραμμα δεν αφήσει περιθώρια για διαβολεύσεις και συνένεση γίνεται μια αναφορά σε ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και αντί να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες προτάσεις μας λέτε ατιοδικία για τη συμμετοχή των κοινικών στα διοικητικά συμβούλια. Kostatinka, du hast jetzt die Zeit ums Doppelte überzogen. Äh, dass das ausgerechnet bei meiner Fraktion passiert, ist nicht in Ordnung. Κωνσταντίνκα, έχεις ολοκληρώσει έχει διπλασιάσει. Παρακαλώ, ολοκλήρωσε. Είναι ένα μη ισορροπημένο σχέδιο. Πιστεύετε πραγματικά πως τα μέτρα που προτείνετε αρκούν για την άρση της περιτοποίηση των εργαζομένων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα απλά να σας ε, θυμίσω ότι δεν μπορεί ο καθένας ε, να μιλάει το διπλάσιο χρόνο από αυτόν που του έχει δοθεί. Δύο λεπτά για τον καθένα και αυτό ισχύει και για τη δική μου πολιτική ομάδα. Κυρία Τάισεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχάς, ε, κυρία Κούνεβα, Μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις όσον αφορά τον ε, κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Αν διαβάσετε το πρόγραμμα του 2016 θα διαπιστώσετε ότι αυτό είναι το πιο κοινωνικό πρόγραμμα που είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε εισάγει την κοινωνική διάσταση στο πρόγραμμα εργασίας και χαίρομαι που το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από το σύνολο του σώματος των ε, επιτρόπων. Επίσης, ε, αν θέλουμε νέες και καλές θέσεις εργασίας, ε, χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη και αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την ε, κοινωνική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση. Χρειαζόμαστε μια μακροοικονομική πολιτική όπου να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες, το σύνολο της κοινωνίας, οι επενδυτές επίσης και έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και στόχος ε, είναι 315 δισεκατομμύρια ευρώ να ε, χρησιμοποιηθούν ε, στην οικονομία. Θα πρόκειται για ιδιωτικούς πόρους που θα κινητοποιήσουν την οικονομία. Έχουμε το πακέτο επενδύσεων που στόχο έχει να δημιουργήσει ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε η αγορά εργασίας να λειτουργεί σωστά. Οι εργαζόμενοι να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους εργαζόμενους, ε, να τους ε, και να τους προστατεύσουμε όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο ήταν ε, να δώσουμε νέα όθηση σε αυτόν. Είχαμε συνάντηση με Ευρωπαίους και εθνικούς ενδιαφερομένους για να δούμε πώς μπορούμε να το οργανώσουμε αυτό με καλύτερο τρόπο στο μέλλον και να του ξαναδώσουμε τη θέση που του αρμόζει. Έχουμε την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Δίνουμε στους ενδιαφερομένους στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τους ζητούμε να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα και τις εθνικές εκθέσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το πρόγραμμα στο σύνολό του και πιστεύω ότι Εάν το κάνετε αυτό θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα ε, κοινωνικά και εργασιακά θέματα ε, χαίρουν πολύ περισσότερη προσοχή από ό,τι συνήθω. Η Λόρα Τζέα, παρακαλώ. Ε, Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα, <coughs> κυρία Επίτροπε. Ενάμισης χρόνος έχει περάσει από τότε που ε, ασχολείστε με αυτό το θέμα και ε, νομίζω ότι από τότε έχει διαφανεί ότι το μόνο που μπορούμε, ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να εφησυχάζουμε. Μας έχετε δώσει κάποια ε, αριθμητικά στοιχεία για την οικονομία μας, μακροοικονομικά, αν δει ε, κανείς την κατάσταση σε επίπεδο μικροοικονομίας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Εκατομμύρια μακροχρόνια άνερθη. Αυτό πραγματικά μας δείχνει ότι έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας ε, και ε, δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση. Η κατάσταση είναι απολύτως ανησυχητική και αυτό σημαίνει ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας πολύ δύσκολη μας μιλήσατε για ένα πρόγραμμα εργασίας μελλοντικό, ενίσχυσης των μακροχρόνια ανέργων. Ε, ο συνάδελφος Μίτοταν ήρθε να μας μιλήσει, μας ε, αναφέρθηκε ακριβώς σε μια εγγύηση παρόμοια με την εγγύηση των νέων για τους μακροχρόνια άνεργους. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ήταν παταγώδηση η αποτυχία της εγγύησης για τους νέους σε διάφορα κράτη-μέλη Ίσως έχετε και εσείς τα ίδια ερωτηματικά. Ε, και εσείς ε, μας είπατε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαχείριση της εγγύησης αυτής για τους νέους ε, ήταν πραγματικά μεγάλη αποτυχία και χάθηκε μια ευκαιρία για τους νέους. Αν λοιπόν ξαναγίνει το ίδιο πράγμα για τους μακροχρόνια άνεργους, μήπως θα γίνει και πάλι το ίδιο πράγμα και θα έχουμε μια ακόμη παταγώδη αποτυχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Αγκαία για την ε, ερώτηση σας αυτής. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι ε, μεγάλο πρόβλημα η ενεργεία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία. Δεν θα μ' ακούσετε να λέω κάτι διαφορετικό. Αυτοί οι δύο πυλώνες συνδέονται και πρέπει ε, ως, ως συνδεδεμένους να τους αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, Η εγγύηση για την εργασία των νέων ε, και τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη, διαρθρωτικές αλλαγές ε, στις οποίες ε, προέβησαν τα κράτη-μέλη, έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς. Εσείς μας είπατε ότι μειώνεται η ανεργία των νέων. Εντάξει, είναι ακόμη σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον κάποια βελτίωση υπάρχει. Θα, ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν κάποιες στατιστικές, το γνωρίζουν αυτό, συλλέγουν ήδη τα στοιχεία αυτά, παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη της εγγύησης για τους νέους. Ε, υπάρχει Υπάρχουν 3,2 δισεκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν και εμείς ελέγχουμε όχι μόνο αν έχουν, διατεθ, αν έχουν αξιοποιηθεί τα ποσά, αλλά ποια είναι και τα αποτελέσματα, πώς έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα και ποια, αποτέλεσμα έχουν, ποια αποτελέσματα έχουν επιφέρει. Θα συλλεγούν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και θα δούμε κατά πόσο οι συστάσεις ε, και οι αλλαγές που ζητούμε από τα κράτη-μέλη είναι επαρκείς, και αν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν αυτή είναι σωστή απάντηση στην, στο ερώτημά μας ή αν πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρώτα όμως πρέπει να δούμε τα δεδομένα, να τα αξιολογήσουμε και μετά θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Τώρα κοιτάξτε, δεν έχουμε ένα κοινωνικό πλωστάσιο επιχειρημάτων να στραφούμε ε, στην ε, δημοσιονομική αρχή για να ζητήσουμε άπειρα ε, ποσά για την ανεργία των νέων. Όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία, έχουμε δει ότι το ίμιση των ανέργων στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι μακροχρόνια άνεργοι. Άνθρωποι δηλαδή που αναζητούν πάνω από ένα χρόνο ενεργά στην αγορά εργασίας μία θέση απασχόλησης. Και αυτό ισχύει. 50% των ανέργων ε, και στη χώρα σας είναι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι χαμηλότεροι οι απόλυτες, είναι χαμηλότερες οι απόλυτες τιμές ενδεχομένως ε, για κάποιες χώρες από ό,τι σε κάποιες άλλες, όμως γενικά το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ζητήσαμε και από τα κράτη-μέλη, κάναμε αυτή τη σύσταση στα κράτη-μέλη να προβούν σε τρία στάδια μέτρων ε, για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καταρχάς, πρέπει να καταχωρηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι. Να σας πω την αλήθεια, αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά πολλά κρατημέλη δεν το κάνουν. Στη συνέχεια, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι πρέπει να κάνουν μια προσωπική αξιολόγηση για να βλέπουμε ποια, ποιο είναι το πρόβλημά τους. Είναι, το πρόβλημα, ας πούμε, ε, της γλώσσας, είναι πρόβλημα μεταφοράς ε, δικαιωμάτων. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είναι λοιπόν μια μεμονωμένη αξιολόγηση των εργαζομένων, των ανέργων, συγγνώμη. Ε, ε πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες. Όταν υπάρχει μια, ένα ενιαίο ε, σημείο επαφής, ε, είναι ευκολότερα. Δεν είναι κάτι, τα πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο έπεσε απλώς από τον ουρανό. Είναι μία πρόταση την οποία υποβάλαμε πριν από μερικούς μήνες. Αυτή τη στιγμή συζητείται στο ΕΠΣΚΟ και ελπίζω ότι Κάτα το μήνα Δεκέμβρη θα εγκριθεί και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Τα κράτη-μέλη βεβαίως πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά ε, ταμεία για να, μπορέσουμε να, να μπορέσουν να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους επανένταξης των ε, μακροχρόνια ανεργών. Ευχαριστώ. Τελευταίο συντονιστής, Ντομινίκ Μαρτά. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Ε, πραγματικά με δυσαρέσκεια λέω ότι ε, πραγματικά ε, ε λέμε Λέμε συνεχώς ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, ε, με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να ε, ικανοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τις, ε, τον εαυτό μας, αλλά πραγματικά αυτό είναι καλό για το ηθικό μας. Όμως αυξάνεται συνεχώς και το ποσοστό της ανεργίας, αλλά και των φτωχών. Το ερώτημά μου όμως δεν αφορά αυτό. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι μέχρι το 2017 θέλει να υποδεχθεί 2 με 3 εκατομμύρια προσφύγων και το το ερώτημά μου είναι το εξή. και είναι και πολύ απλό. Πώς και με τι χρήματα έχετε σκοπό να βρείτε δουλειά σε αυτούς τους πρόσφυγες, ε, πώς και με τι χρήματα έχετε σκοπό να διαχειριστείτε το, τα συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα των οικογενειών αυτών χωρίς αυτό να είναι εις βάρος των ε, πολιτών των κρατών μελών. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που κάναμε εξ αρχής όταν είδαμε ότι η κρίση των προσφύγων ήταν πολύ ε, μεγάλη, όταν δηλαδή το θέμα των προσφύγων ε, έγινε κρίση, πλέον, έγινε πλέον μια κρίση. Ζήτησα από όλους να ε, βρεθούμε εδώ ε, στις Βρυξέλλες για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε κοινωνικός και οικονομικός ε, αυτούς τους πρόσφυγες που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα όλων αυτών των δικαιωμάτων της ε, διεθνούς προστασίας. Αυτό που ζήτησα λοιπόν ε, στις διάφορες υπηρεσίες αλλά και ε, στους διευθυντές των υπηρεσιών των κρατών μελών είναι να μας πούν πώς μπορούν να κινηθούν, αν μπορούν να κινητοποιήσουν προγράμματα και να υποβάλουν προτάσεις τροποποίησης, ότι θα είμαστε ευέλικτοι, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε στις πλάτες ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό. Για όλα τα υπόλοιπα μπορώ να σας καθησυχάσω και να σας διαβεβαιώσω ότι ο στόχος μας ε, δεν είναι να ε, κάνουμε σύγκληση προς τα κάτω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και έχει επιβεβαιωθεί και από το Διεθνές Ταμείο και από τον ΟΣΑ ότι όταν η σύγκληση οικονομική και κοινωνική είναι πολύ μεγάλη σε ένα κράτος μέλος ή μεταξύ των κρατών μελών, αυτό δεν είναι καλό για την οικονομική ανάπτυξη. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη ε, σύγκληση, χρειαζόμαστε ε, ισότητα ευκαιριών για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και για να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε, αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό αναφέρεται σαφέστατα και θα το δείτε αυτό όταν θα διαβάζετε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε να υπάρξει μια σύγκληση προς τα πάνω και καθόλου προς τα κάτω. Σε καμία περίπτωση υπήρξε οικονομική κρίση ε, η οποία βέβαια μας έθεσε σε μια διαφορετική αφετηρία και αυτό το συνειδητοποιούμε. Ε, είμαστε στο πλαίσιο μιας ε, οικονομικής ε, μεταρρύθμισης, υπάρχει και η παγκοσμιοποίηση, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι με αυτό, αλλά είναι μια εξέλιξη της ανθρωπότητας που δεν, ε, στην οποία δεν μπορούμε να αντιταχθούμε, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να τη συνοδεύσουμε, πρέπει να την αποδεχθούμε και να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες ε, σε όλους. Αυτό είναι ο στόχος μας και είναι αυτό το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ θερμά. Και τώρα φτάνουμε στην ανοιχτή συζήτηση. Έχουμε 16 ομιλητές στον κατάλογο. Υποθέτω ότι μπορούμε τώρα να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Και δεύτερη ανακοίνωση. Προτείνει να πάρει το λόγο για ένα λεπτό ο καθένας, ώστε να έχουμε έστω και μια ελπίδα ότι θα ακούσουμε την απάντηση της ε, κυρίας ε, Τάισεν, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξή μας. Ε, ούτε και εδώ βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Η Μαρίτα και έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που η κυρία πίτροπος τηρεί την υπόσχεση του κυρίου Ιούνκερ που ήταν η ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά και όχι κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν μπορούμε να, ανταγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε με άλλα μέρη του κόσμου εάν είμαστε πιο φτηνοί. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο ευφυείς. Το κοινωνικό ντάμπινγκ δεν είναι η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ωστόσο, ανησυχώ. διότι πιστεύω ότι η αρχή της ίσης αμοιβή θα πρέπει να ε, λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, την Συμφωνία ΤΙΣΑ έχουμε πρόβλημα κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αλλάξουμε αυτό. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Ανησυχώ λοιπόν για το τι θα γίνει εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λύσει πρώτα τα δικά της προβλήματα προτού ανοίξει τις αγορές της ε, απέναντι σε ε, παράγοντες ε, τρίτων χωρών. Ποια είναι η θέση της Επιτρόπου για το θέμα αυτό και πότε θα έχουμε τα πραγματικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση του, του κοινωνικού ντάμπινγκ. Πάντως έχετε την απόλυτη υποστήριξη τη πολιτική μου Ο Όλε Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο που είναι παρούσα εδώ στην Επιτροπή μας. Χάρηκα που άκουσα την ε, παρατήρησή τη ε, για την ε, ασφάλεια και την υγιεινή και ιδιαίτερα όσον αφορά τις καρκινογόνες ουσίες. Σίγουρα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ελπίζω η Κομισιόν επίσης να έχει μια φιλοδόξη στρατηγική από το 2014 μέχρι το 2020 και λίγο με ανησυχεί όταν ακούω για απλοποίηση λιγότερες οδηγίες, πώς αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Ελπίζω η Κομισιόν να επιμένει σε μια φιλόδοξη στρατηγική από πλευρά τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Τάισεν που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας για να συζητήσετε μαζί μας. Αναφέρατε κάποιες προτάσεις που ήδη έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μάλλον ήπια όμως πολλά από τα μέσα αυτά. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία για την ανεργία, η ε, γονική άδεια, και η πρωτοβουλία για την ε, ισορροπία ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Η ερώτησή μου είναι, εάν θέλουμε να λύσουμε αυτήν ε, την σκληρή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χρειαστούμε περισσότερε νομοθετικέ προτάσει με ισχυρή συμμετοχή, ιδιαίτερα τη Επιτροπή μα, αλλά και γενικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να λύσουμε τι προκλήσει, για να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξή. Επιθανότατα να γνωρίζετε ότι σήμερα είναι η μέρα των ασκούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε προωθήσει ε, ένα πλαίσιο ποιότητα για τι θέσει ασκούμενων και ε, θα λάβουμε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας στο τέλος της χρονιάς. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να αυξήσετε την ποιότητα των ε, θέσεων ασκούμενων εντός Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την παρουσία σας και το πρόγραμμά σας. Ε, πολλές ερωτήσεις έχω. Μιλήσατε για την κοινωνική σύγκληση. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει κοινωνική απόκληση. Ισχυρή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε η εκπρόσωπός μας έναντι των άλλων επιτρόπων, ούτως ώστε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος όλα τα μέτρα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κρίση για όλε τι χώρε που δεν έχουν φτάσει σε ένα μήνυμα επίπεδο. Είπατε ότι πρέπει να υπάρξει καινοτομία, κατάρτιση, ψηφιακά και επίκειται η COP21. Δεν μιλήσατε για τι πράσινε θέσει εργασία, ούτω ώστε να είμαστε ηγέτε στην προστασία του περιβάλλοντο παγκόσμια. Ποιο είναι το πρόγραμμά σα για αυτέ τι πράσινε θέσει εργασία. Τρίτον, συνδυασμό ε, ιδιωτικού και πραγματικού βίου. Ξέρετε ότι η άδεια μητρότητα ήταν έτοιμά μα να αναθεωρηθεί δηλαδή η οδηγία. Όμως δεν έγινε. Λόγω του refit. Δεν βλέπουμε ούτε καν οδικό χάρτη. Ή μάλλον ο οδικός χάρτης δεν επαρκεί. Και τελευταίο. Η κινητικότητα. Αλλά η κινητικότητα δεν είναι μόνο η απόσπαση. Η απόσπαση είναι μόνο το τμήμα της κινητικότητας. Φυσικά είναι σημαντική η κινητικότητα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούν την απόσπαση οι επιχειρήσεις είναι για να παρακάμψουν ε, το σύστημα προστασίας των εργαζομένων. Πρέπει λοιπόν να τους αφαιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ελιζαμπέτ ε, Νοέν Σαρτιέ. Ευχαριστώ. Τρία θέματα θα θίξω. Πρώτον, η κατάρτιση των εργαζομένων θέλω να υπάρξει επανάσταση από αυτού. Επιτέλους, να βοηθήσουμε να αποκτούν δεξιότητες και όχι απλώς τυπικά προσόντα και διπλώματα. Να έχουν ουσιώδεις δεξιότητες για να μπορέσουν όντως να βρουν εργασία. Άρα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος κατάρτισης, να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης της κατάρτισης και να εξελιχθεί ο κοινωνικός διάλογος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, Μιλήσατε για τις εγγύησεις ε, για την εργασία των νέων. Αλλά δεν προχωράει αρκετά γρήγορα αυτό. Εσείς ήσασταν ε, η κύρια προθετική δύναμη γι' αυτό όταν θέλαμε αυτή η πρωτοβουλία για τους νέους να περάσει από 1 σε 30% προχρηματοδότησης. Να εργαζόσαστε, να εργαστείτε περαιτέρω γι' αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε σύντομα για παράδειγμα όλη αυτή η συλλογή στοιχείων και τα λοιπά όλες αυτές οι καθυστερήσει. Πρέπει πραγματικά να πιέσουμε αφόρητα τα κράτη-μέλη για να επιταχύνουν και εμείς να επιταχύνουμε. Και τρίτον, άδεια μητρότητα. Τέσσερα σημεία περιέχει η κατάρτιση των νέων γυναικών, οι αμοιβέ του, οι σταδιοδρομίες του και η φτώχεια που θίγει τι γυναίκε και ε, το, η άδεια μητρότητας αφορά και τα τέσσερα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να ε, τηρήσουμε το χρόνο μας και είμαι επισμένος ότι η Τανούτα θα τον τηρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, ε, κύριε Επίτροπε. Μακάρι να τα λέγαμε πιο συχνά εδώ γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι ανταλλαγές απόψεων μαζί σα. Αναφερθήκατε στους κοινωνικού εταίρου. το διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Νομίζω ότι ο συνεχής και βιώσιμο διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών είναι πολύ σημαντικό. ιδιαίτερα στα πλαίσια τη απόσπαση των εργαζομένων. Αλλά και για άλλε διάφορε ευέλικτε μορφέ απασχόληση. γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εξελίξει στην οικονομία συμβαδίζουν με την εξελίξη στην προστασία, με τη διατήρηση τη προστασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει εταιρική σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι η ραχοκοκαλιά για την επιτυχία μα. Πώ θα πείσουμε του εργοδότε να παίζουν πολύ ενεργό ρόλο. Δεν είναι ισότιμο αυτό ο διάλογο όπω γίνεται τώρα. Τι θα κάνουμε ούτω ώστε να συμμετέχουν όλοι ισότιμα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Άλλη ερώτηση. Τι θα κάνει η Κομισιόν ούτω ώστε να τονίσει περισσότερο ότι πρέπει να ελέγχεται ο τρόπος απορρόφησης πόρων από τα κοινωνικά ταμεία ούτω ώστε να διασφαλιστεί στενότερη σχέση μεταξύ των εταιριών και τη εκπαίδευση, δηλαδή μεταξύ της εργασία και τη εκπαίδευση, ούτω ώστε οι δεξιότητε των εργαζομένων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και αυτό που δημιουργούν νέε εργασίες Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο πρόεδρο Σβέν Κύριε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα, εβδομάδα ήμουν στην πράσινη εβδομάδα στην ε, περιοχή μου, τη Σαξονία Άνχαλτ. Εκεί έχουμε υψηλή ανεργία. Δεν έχει ολόκληρη η Γερμανία χαμηλή ανεργία. Ορισμένα τμήματα τη Γερμανία έχουν υψηλή. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μίλησαν μαζί μου και μου είπαν ότι προσπαθούν να δώσουν εργασία σε πρόσφυγες, αλλά πολλοί δεν έχουν καθόλου προσόντα μέχρι 30% είναι αναλφάβητη. Συγκεκριμένη ερώτηση. Τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνει η Επιτροπή για να δοθούν περαιτέρω πόροι, ούτως ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για να δώσουν θέσεις εργασίας στους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θαυμάσια τηρήσατε και το χρόνο σας. ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανακοίνωση για την ε, ύπαρξη νέας ουσίας ε, στην ε, απόσπαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Αυτό ακριβώς θέλουμε και αναμένουμε εναγωνίως τις προτάσεις σας. Την απάντησή σας στην κυρία Μάικιντάρ περί απόσπασης δεν ήταν αυτό ακριβώς που περίμενα. Το να εφαρμοστεί η οδηγία δεν είναι επαρκές. Χρειαζόμαστε πραγματική δράση επί της οδηγίας και χάρηκα που το είπατε αυτό σαφώς σαφέστατα. Πραγματικά με πολύ χαρά περιμένουμε τις ε, προτάσεις σας σύντομα. Ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης μας είπε ότι δεν υπάρχει επισφαλής εργασία, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επισφαλούς εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ε, σωστό και θα ήταν καλό να τα ακούσουμε και από το δικό σας στόμα και όσον αφορά το ότι ε, είπατε ε, ότι η ανεργία στην Ισπανία και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ε, υψηλή. Μπορείτε να μας απαντήσετε και στη δύσκολη ερώτηση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας γιατί βλέποντας την κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να διαχειρίζεται τα ζητήματα και να τα εγγράφει ε, σε ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο. Χάρηκα με αυτά που μας είπατε για την οδηγία περί απόσπασης, η αναθεώρηση και η επανεξέταση είναι δύο διαφορετικά πράγματα η αναθεώρηση είναι μια νομοθετική προσέγγιση και έχω το εξής ερώτημα. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι αν, ε, ε, ε, υπάρχουν διακρίσεις στο, στην αγορά εργασίας, δεν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ίση αμοιβή στον ίσο τόπο εργασίας ε, και αυτό να είναι εις βάρος της ε, ίσης ε, κοινωνικής προστασίας. Δεύτερον, πρέπει να δούμε και το κοινωνικό πυλώνα. Πάρα πολύ καλά κάνατε που το αναφέρατε αυτό, αυτό τόσες πολλές φορές αν ε, ακολουθήσουμε την υφιστάμενη ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, γιατί βλέπουμε ότι η απόκληση ε, ήταν το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου και όχι τόσο η σύγκληση, πώς θα μπορέσουμε να, δώσουμε, να, να, να υπάρξει εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο κοινωνικό πυλώνα, όταν λέτε ότι υπάρχει, θέλουμε να υπάρχει σύγκληση προ τα πάνω και όχι προ τα κάτω. Μήπω υπάρχει μια παγίδα σε αυτό. Η Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε να μας συναντήσει σήμερα το πρωί. Απαντήσατε ήδη σε αρκετές ερωτήσεις. Θα ήθελα να συμμεριστώ την άποψή σας ως προς την αναγκαιότητα να υπάρξει μια νέα στρατηγική για νέες ε, δεξιότητες. Είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική πρόκληση, ε, ειδικότερα στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, την οποία θέλουμε να ε, αναπτύξουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νέες δεξιότητες σημαίνει βέβαια νέα ε, εκπαίδευση και νέα διπλώματα. Σήμερα όμως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολίτες των κρατών μελών ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίε για την αναγνώριση και την επικύρωση ε, των σπουδών που ε, κάνουν στο εξωτερικό. Και αυτό πραγματικά παρεμποδίζει την κινητικότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς μεγαλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων. Η κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε, κυρία Επίτροπε πάρα πολύ καλό το πρόγραμμά σας ε, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενισχυμένη συνεργασία που ε, υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου είναι και πάλι η σύγκληση και πιο συγκεκριμένα είναι πώς ε, έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το επόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την ενίσχυση της σύγκλησης. Τρία βασικά σημεία. Οι στόχοι, γιατί οι στόχοι πρέπει να καλύπτουν και τις κοινωνικές ανισότητες. Δεύτερον, οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα, γιατί και αυτές θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν και το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Και το τρίτο θέμα είναι η οικονομική υποστήριξη, γιατί βέβαια τα κοινωνικά ταμεία μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα, να αξιοποιήσουμε την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και νομίζω ότι πέρα από αυτό θα ε, χρειαστεί μια πραγματική ε, δημοσιονομική ε, ικανότητα των χωρών της Ευρωζώνης. Η κυρία Μπλινκοβιτσιούτε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή μας ενέκρινε πρόσφατα μία έκθεση σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας και καλέσαμε στην έκθεσή μας αυτής, αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει μία εγγύηση για τα παιδιά, να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι κάθε παιδί που ε, ζει στη φτώχεια θα έπρεπε να έχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη, γεύματα και εκπαίδευση και νομίζω ότι αυτή η εγγυήση θα μπορούσαν να, να μας βοηθήσει να λύσουμε πολλά προβλήματα που θα εμφανιστούν μεταγενέστερα μεταξύ των οποίων η ανεργία και έτσι μπορούμε να σταματήσουμε τον κύκλο της φτώχειας. Συμφωνούμε... Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία προσπαθώντας να αναθεωρήσουμε την στρατηγική για το 2020, όπου ένας από τους στόχους μας ήταν η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Γι' αυτό νομίζω ότι θα είχε νόημα να υπάρξει αυτή η εγγύηση τώρα. Επίσης, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της επισφαλούς εργασίας. Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τι θα προτείνει στα ε, κράτη-μέλη ώστε να ε, εξαλειφθεί το πρόβλημα της επισφαλούς εργασίας. Επίσης είπατε ότι θα υπάρξει μία οδηγία για την άδεια ε, προκειμένου να φροντίσει κανείς ε, σοβαρή ασθένεια εντός του ε, οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πότε μπορούμε να περιμένουμε αυτήν την οδηγία. Ευχαριστώ ο αθέμητος ανταγωνισμός ε, αυτή τη στιγμή υπονομεύει την ε, εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαφές. Μιλήσατε για την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων και την ομολογία του δικαστηρίου που συχνά ε, δεν είναι πολύ ευνοϊκή για τους εργαζομένους. Σήμερα η οδηγία της απόσπασης και η νομική βάση δεν έχει να κάνει με το άρθρο 153 της συνθήκης αλλά με άρθρα τα οποία που αφορούν την ε, είσοδο ε, στην ε, αγορά. Μήπως θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν η νομική βάση σήμερα της οδηγίας περί απόσπασης προκειμένου να ε, ισχύς της εφαρμογής της να είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα. Ο Τόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Επίτροπε, κάποιοι συνάδελφοι παραπονέθηκαν για τη δουλειά της ε, Κομισιόν, αλλά εγώ το βλέπω διαφορετικά. Βλέπω ότι έχετε φιλόδοξο θεματολόγιο και ε, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε τη φετινή χρονιά με προηγούμενες. Ε, τα κράτη-μέλη όμως δεν είναι διατεθειμένα να επιδείξουν αλληλεγγύη, για παράδειγμα ε, όσον αφορά τους ε, πρόσφυγες. Είναι λάθος αυτή η οδός. Όσον αφορά την εγγύηση για, την, για τους νέους. Πιστεύω ότι αποτελεί καλή βάση. Και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μακροχρόνια ανεργία. Δεν θα πρέπει όμως να συνδυάσουμε τα θέματα μεταξύ τους, ε, δηλαδή την προστασία των ανθρώπων ε, με την ε, ανεργία. Θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν αγνοούμε τα θέματα αυτά και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την άρνηση του κόσμου να τα συζητήσει. Ευχαριστώ. Ο κ. Λοπέζ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που ήρθε εδώ και μας μίλησε για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη, για τις κοινωνικές ανισότητες που θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με τον κοινωνικό πυλώνα. Βεβαίως ξέρουμε τι επιρροή, τι, πόσο θίγουν την οικονομία μας και γενικότερα το ευρωπαϊκό όραμα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τους θύλακες φτώχειας που έχουμε, την αργία των νέων, αλλά υπάρχουν και άλλοι θύλακες φτώχειας. Για παράδειγμα η παιδική εργασία τρομερό δυναμητίζει ε, την αξιοκρατία που θεωρούμε ότι είναι η βάση της οικονομίας μας, η βάση της κοινωνίας μας. Πώς είναι δυνατόν να δεχόμεθα κάτι τέτοιο. Πολλά από τα προγράμματά μας σχετίζονται όμως με τους ε, μηχανισμούς λήψης σκληρών αποφάσεων, όπως το εξάμεινο. Πώς θα εισαγάγουμε στα πλαίσια της προσπάθειας οικονομικού συντονισμού τα θέματά μας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, πολύ σύντομα, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα με βάση την κατάρτιση και προετοιμασία. Συμφωνώ με αυτά που είπατε, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε κάνει το αντίθετο. Έχει γίνει εσωτερική υποτίμηση σε πολλές χώρες. Έχει καταρρεύσει η αγορά εργασίας. Όλα αυτά επειδή είμαστε δεμένοι με το ευρώ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι αντιφατικά. Ευχαριστώ. Η Άννα ο Άρνολτ Γκέρκερ. Βεβαίως η αμοιβή, αλλά ε, τι έννοια έχει αυτή η παιδική, ή συγγνώμη, η, η γονική ή η μητρική άδεια. Ξέρετε ότι πολλοί εργάζονται όλο το χρόνο και δεν έχουν καμία δυνατότητα να πάρουν ε, άδεια. Και εάν οι εργαζόμενοι δεν έχουν επαρκείς πόρους, τότε υπάρχει φτώχεια και για τα παιδιά. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στην Επιτροπή μας. Πόσο επιτέθηκαν οι συντηρητικοί κατά της ε, οδηγίας ε, για την άδεια μητρότητας. Ενώ οι συνάδελφοι από την αριστερά ήθελαν να τα βάλουν όλα μέσα σε αυτή την οδηγία, ούτω ώστε να μην μπορεί πλέον να εφαρμοστεί. Για λόγους ιδεολογικούς γίνονται όλα αυτά. Το Συμβούλιο μετά λοιπόν την απέρριψε. Εγώ ως Ευρωβουλευτής του κόμματος για τις οικογένειες από την αρχή της ε, νομοθετικής αυτής περίοδου είπα ότι χρειαζόμαστε λειτουργική προστασία της μητρότητας. Θέλουμε μία νέα μορφή της αντίστοιχης οδηγίας. Κυρία Επίτροπε, θεωρώ ότι έχω δίκιο γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορετική αμοιβή για την ίδια εργασία. Θέλουμε λοιπόν να λειτουργούν οι κανόνες μας. Πρέπει να δίδεται σε όλη την Ευρώπη μία αμοιβή για τους γονείς και μία ελάχιστη αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους και να υπάρχουν επαρκείς βρεφονιπιακοί σταθμοί γιατί πολλοί γονείς και πολλά παιδιά λείπουν από τις κοινωνίες μας. Ολοκληρώσαμε έτσι τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών, δεν σας ζηλεύω που θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις μέσα σε 15 λεπτά. Η Επίτροπος, ε, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Καταρχάς, ε, όσον αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πιστεύω ότι η πιο σημαντική ερώτηση ήταν πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με μία νομοθετική πράξη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία πολιτική εγκάρσια θα πρέπει να εξετάσουμε τα ελάχιστα δικαιώματα που θα πρέπει να έχει κανείς και κατόπιν θα πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να συνάψουν συμφωνίες για τα σημαντικά θέματα. και να συζητήσουμε τα κεντρικά θέματα για να δώσουμε σάρκα και οστά στην πολιτική αυτή. Μπορούμε, πιστεύω, να το κάνουμε αυτό. Και η διασυνοριακή πτυχή αποτελεί ε, μέρος ε, του πακέτου ε, για την απασχόληση. Κύριε Κρίστενσεν, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας σχετικά με για τις καρκινογόνες ουσίες. Θα εξετάσουμε το θέμα αυτό κατά την αναθεώρηση του συνολικού πακέτου για την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τις καρκινογόνες ουσίες και θα το κάνουμε μόλις έχουμε στα χέρια μας τα απαραίτητα στοιχεία. Κυρία Ρένκε, όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ανεργία, είπατε ότι είναι ήπια η προσέγγιση μα στον τομέα αυτών. Φυσικά θα ήθελα να υπάρχει δεσμευτική νομοθεσία στον τομέα αυτών. Θα ήθελα πολύ να υποβάλω στο Κοινοβούλιο σχέδιο νομοθεσίας. Ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Θα πρέπει να εργαστούμε με βάση αυτά που έχουμε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο περιφερειακό, τοπικό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα, διότι όσο μεγαλύτερο διάστημα παραμένει κανείς άνεργος, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει μια θέση απασχόλησης. Χρειαζόμαστε το εργατικό δυναμικό. Θα του χρειαστούμε στο μέλλον του ανθρώπου αυτού και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε ανθρώπους κοινωνικά απεκλεισμένους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια καλά δομημένη προσέγγιση στα θέματα αυτά, ώστε να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην ε, αγορά εργασίας. Ε, χρησιμοποιούμε τις εξουσίες μας στο βαθμό που μπορούμε. Κατόπιν έχουμε το θέμα της ισορροπίας ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Ε, και εδώ έχουμε ήπια προσέγγιση. Είχαμε υποβάλει σχετική νομοθεσία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα ήταν ε, καλή πολιτική να εφαρμόσουμε αυτά που προτείναμε το 2008. Εάν ε, δεν υπάρχει βούληση να ακολουθήσουμε την οδό αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. θα πρέπει να θεωρήσουμε την απόσυρση της οδηγίας για, τη μητρική, ε, για την άδεια μητρότητα σε θετικό βήμα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις έγκυες στον χώρο εργασίας και θα πρέπει να φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε και τους πατέρες στο πακέτο αυτό. Θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες και θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά όχι μόνο ε, για του γονεί, ε, για την περίπτωση των παιδιών δηλαδή, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα. Θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα κοινωνική και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ακριβώς ε, γι' αυτό ε, έχουμε... Εργαζόμαστε πάνω σε ένα συνολικό πακέτο. Επίσης, όσον αφορά τις θέσεις ασκούμενων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικό θέμα στο θεματολόγιο μας και νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβατε και από την εισαγωγή που έκανα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε τις δεξιότητες και την αναγνώριση των δεξιοτήτων. Στόχος εδώ είναι να φροντίσουμε οι δεξιότητες να είναι όσο γίνεται πιο διαφανείς και αναγνωρίσιμες. Και αυτό θα πρέπει να γίνει διασυνοριακά. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις θέσεις ασκούμενων, έχουμε προωθήσει το θέμα αυτό Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε να υπάρχουν επαρκείς θέσεις ασκούμενων. Ξέρουμε ότι είναι καλό σύστημα και θέλουμε να συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κατάλληλο πλαίσιο και θέλουμε τα κράτη-μέλη να μαθαίνουν το ένα από το άλλο. Θέλουμε επίσης να εισάγουμε το σύστημα αυτό στα κράτη-μέλη που δεν γνωρίζουν ένα τέτοιο σύστημα. Μιλήσαμε για την κοινωνική σύγκληση. Κύριε Αρένα, αναφερθήκατε στις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Και είπατε ότι δεν το καλύψαμε. Έχετε δίκιο. Μιλάμε συνέχεια για ψηφιακέ θέσει απασχόληση, αλλά και η πράσινη οικονομία είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να τη στηρίξουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ανάπτυξη, ώστε να υπάρχουν και εκεί ευκαιρίες απασχόλησης. Και όσον αφορά το θέμα της άδεια μητρότητας, χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω και με αυτό το θέμα. Πρέπει να εξετάσουμε τις ανάγκες και να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το καλύτερο δυνατό μέσο. Χαίρομαι που στηρίζεται το θέμα της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και αναγνωρίζεται ότι δεν είναι απλά θέμα εφαρμογής του νόμου. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της χώρας προέλευσης ε, και της χώρας υποδοχής. Βρέθηκα την Ντανούτα στην Κρακοβία για τις ημέρες μελέτης πάνω στο θέμα αυτό. Στην Πολωνία οι άνθρωποι επιθεωρητές ανησυχούν πολύ σχετικά με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στο κράτος μέλος αναγνώρισης, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εφαρμοστική οδηγία για να διασφαλίσουμε την πρόοδο στον τομέα αυτών. Και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων. θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των εργοδοτών στο πακέτο. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν τα απαραίτητα μέσα ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή εκπροσώπηση. και να ληφθούν μέτρα ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε οδηγίες στον τομέα αυτό όσον αφορά την εκπαίδευση και τις δεξιότητε. πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε για τη συμμετοχή των εργοδοτών και θα πρέπει να έχουμε πιο στενές επαφές με τον επιχειρηματικό κόσμο Θα πρέπει να φροντίσουμε η εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχουμε να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Μιλήσαμε για την μεγάλη ισορροή μεταναστών και προσφύγων στις χώρες μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαθέτει πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των ανθρώπων αυτών και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τους πρόσφυγες. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας, να έχουμε καλύτερο έλεγχο και όπως είπε η κυρία Μωρά, θα πρέπει επιγόντως να αυξήσουμε το ποσοστό προχρηματοδότησης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε αποτελεσματικά στον τομέα αυτών στην Ισπανία και στην Ελλάδα γιατί είναι τόσο υψηλή η ανεργία. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε αυτό επαόριστον. Αλλά νομίζω ότι το θέμα που θα πρέπει να συζητάμε είναι οι προσδοκίες μας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε τη λιτότητα για όλα τα προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιες από τις υποδομές που μπορεί να χωλένουν σε κάποιες χώρες. Κάποιοι τομείς στην Ισπανία ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Μάθαμε από αυτά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αντιμετωπίζουμε στο μέλλον τις μακροοικονομικές ανισορροπίες εγκαίρως. Όσον αφορά τους κοινωνικούς πυλώνες. Έχουμε τον κοινωνικό πυλώνα δικαιωμάτων. γιατί να θεωρούμε ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε σύγκληση προς τα πάνω και όχι σε έναν φαύλο κύκλο. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Έχουμε περισσότερους συμμάχους τώρα στις ε, χώρες της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να συνεργαστούμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν. εάν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό εντό τη ΟΝΕ. Ε, πιστεύω ότι στη δεύτερη φάση θα μπορούμε να είμαστε πιο αυστηροί και να μιλάμε για δεσμευτικού στόχου. Αυτό είναι και ένα από του στόχου. Ε, στο πλαίσιο της ε, εμβάθυνσης ε, της νομισματικής ένωσης. Θα πρέπει <clears throat> να φροντίσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την εσωτερική αγορά και να φροντίσουμε να εργαζόμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση για να ενισχύσουμε τον κοινωνικό πυλώνα θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν καλύτερα κίνητρα στον τομέα αυτών. Επίσης, στέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με την αναγνώριση δεξιοτήτων ε, και επαγγελματικών προσόντων. Απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά στον τομέα αυτών. Δεν είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στο πρόγραμμα όμως θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για περισσότερη και καλύτερη αναγνώριση τίτλων σπουδών. Θέλουμε να το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι, είναι μέρος του πλαισίου δεξιοτήτων και θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα στον τομέα αυτών για να σημειώσουμε πρόοδο. Η κυρία Ροντρίκες και άλλοι μίλησαν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για το πώς Μπορεί να υπάρξει σύγκληση στον κοινωνικό πυλώνα εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ακόμα ασχολούμαστε με το εξάμεινο του 2016. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας, διότι για να γίνει αυτό πρέπει να θέσει κανείς ε, σημεία αναφοράς, benchmarks, και θα πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους μας. Εργαζόμαστε όμως προς τη σωστή κατεύθυνση και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του εξαμήνου. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τη φροντίδα των παιδιών, ε, τις ε, ε, τα επιδόματα εργασίας κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε αυτά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μιλήσαμε επίσης για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Υπάρχει η έκθεση για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά για την Νομισματική Ένωση. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Η παιδική φτώχεια βεβαίως είναι σημαντικό. Η ε, στόχοι της Ευρώπης 2020 περιλαμβάνουν και την καταπολέμηση της ε, παιδικής φτώχειας. Ξέρουμε ότι αντί να μειωθούν κατά 5 εκατομμύρια όπως ε, θέλαμε, όπως είχαμε θέσει ως στόχο, έχουμε δύο παραπάνω. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα μειώνεται λίγο η φτώχεια. Είδαμε ότι από 124 εκατομμύρια μειώθηκε στα 121. Αυτό ε, βεβαίως είναι θετικό, αλλά είναι επίσης λόγος ε, για να ντρεπόμαστε γιατί έχουμε ακόμη λοιπόν 121 εκατομμύρια φτωχών και βεβαίως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, φτώχεια των ε, παιδιών ιδιαίτερα στα πλαίσια χορήγησης καλύτερης πλαισίωση των παιδιών. Εάν υπάρχει καλύτερη πλαισίωση των παιδιών, περισσότερη σταθμή, περισσότερες δυνατότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης, αυτό οπωσδήποτε θα βελτιώσει μακροπρόθεσμα την απασχολησιμότητά τους εάν όλοι οι γονείς και αυτοί που είναι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δυνατότητα καλύτερης πρόβασης στην εργασία λόγω αυτών των συνοδευτικών μέτρων, τότε αυτό σημαίνει ότι δίνουμε μια καλύτερη ευκαιρία σε όλους και τα παιδιά και τους γονείς και καλύτερη εξορρόπηση ε, εργασίας και οικογενειακού βίου και αυτό μειώνει και κατά πολύ τον κίνδυνο τα παιδιά να υποφέρουν αργότερα από την ε, φτώχεια. Ε, μετά τέθηκε το ερώτημα του κ. Μπάλαστ για την νομική βάση για την οδηγία για την απόσπαση. Και υπόθηκε ότι δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η νομική βάση. Έμαθα και νωρίτερα όταν ήμουν ε, εδώ στο Κοινοβούλιο, ότι και, αλλά και τώρα που εργάζομαι στην Κομισιόν, ότι αυτά πρέπει να τα αφήνουμε στους ε, νομομαθείς γιατί είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Αλλά οποτεδήποτε κάνουμε προτάσεις πρέπει οπωσδήποτε να βασίζονται στη σωστή νομική βάση. Και τώρα βεβαίως ο παλιός νάρφος Τόμας ε, Μαν. Ευχαριστώ Τόμας για τις ε, παρατηρήσεις σου, ευχαριστώ για την ε, θετική σου αντίδραση στο πρόγραμμά μας. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι το πρόγραμμα εργασίας είναι φιλόδοξο. Και χαίρομαι που και εσείς προσωπικά αλλά και άλλοι που εκφράστηκαν το τόνισαν αυτό. Χαιρόμεθα γι' αυτό και φυσικά μας ενθαρρύνει για την περαιτέρω εργασία μας. Να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο την κοινωνική διάσταση της οικονομίας μας. Ε, ρωτήθηκε κατόπιν από τον Σνάρφο Λόπεθ πώς θα συμπεριληφθούν τα κοινωνικά θέματα στη γενικότερη εργασία μας. Μα το κάνουμε αυτό. Το επιδιώκουμε, προσπαθούμε να το διασφαλίσουμε μέσω εισαγωγής ε, δικτών για την ε, διαδικασία μακροοικονομικής ισορροπίας. Έχουμε κοινωνικούς δείκτες. Το είπαμε αυτό από την αρχή Ήδη έχουμε επιτύχει να συμπεριληφθούν αυτοί οι κοινωνικοί δείκτες, δείκτες απασχόλησης, ανεργίας κτλ. Και το λαμβάνουμε υπόψη, λοιπόν όπως είπα, για την διαδικασία μακροοικονομικής, μακροοικονομικής ανισορροπίας για τα κράτη-μέλη. Έτσι ούτως ώστε να καθίσταται σαφής η κοινωνική επίπτωση των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται. Επίσης τέθηκε μία ερώτηση για την προστασία της μητρότητας ε, και της γονικής άδειας, ε, ίση αμοιβή, οικογενειακή πολιτική κτλ. Ελπίζω και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτή τη νέα αρχή για την εξορρόπηση εργασίας και οικογενειακού βίου να ληφθούν υπόψη περισσότερο οι ανάγκες των εγγύων και των ε, ε, μητέρων με μικρά παιδιά, αλλά και των ανδρών βεβαίω, των γονέων γενικά με μικρά παιδιά. Υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών. Και πρέπει οπωσδήποτε και οι γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά και οι άλλοι που μόνοι τους ε, βοηθούν άτομα στο οικογενειακό τους περιβάλλον που έχουν ανάγκη προστασίας, όλοι αυτοί και οι μονογονικές οικογένειες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όλοι αυτοί είναι κοινοί μας στόχοι είναι στόχοι που μέσω καλή συνεργασία κατά το 2016 πιστεύω ότι θα του ε, επιτύχουμε σε ένα βαθμό. Πρόεδρο ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. όπω όλοι διαπιστώσατε, η Επιτροπή μα, και εσείς λοιπόν θα διαπιστώσετε κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή μας λοιπόν, η, η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, πάντα θέλει να μάθει περισσότερα από αυτά που θέλει να της πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή που είναι σε θέση να τη πει η Επιτροπή, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη φύση της Επιτροπής μας. Πιστεύω ότι ως Επιτροπή από τη φύση μας θέλουμε κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό από, την, ε, από αυτά που θέλει η Επιτροπή για τα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω ότι αυτά βοηθούν τη συνεργασία μας. Είπατε ότι θέλετε να αυξηθούν ε, οι θέσεις εργασίας. Χαιρόμεθα. Όμως το πρόβλημα είναι ότι με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε αυτές οι νέες θέσεις εργασίας θα είναι επισφαλείς και δεν θα επαρκεί αμοιβή για να ζήσει κανείς από αυτές τις θέσεις εργασίας και κατά τη γνώμη μου και είμαι βαθιά πεπισμένος γι' αυτό δεν λύνουμε το πρόβλημα έτσι γιατί θα πρέπει να συμπληρωθεί λοιπόν το εισόδημα με άλλες κοινωνικές μεταφορές αλλιώς θα έχουμε σοβαρά προβλήματα άρα μακροπρόθεσμα δεν λύνεται το πρόβλημα. Μακροπρόθεσμα στόχο μα πρέπει να είναι να δημιουργηθούν υψηλού επίπεδου θέσει εργασία. Και αυτό θα το πούν και οι τρει νομίζω ε, θεσμοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ και ελπίζουμε τώρα να λάβετε υπόψη αυτά που σας είπαμε στη συνέχεια της εργασίας σας. Έχουμε χρόνο για ε, δεν έχουμε χρόνο για διάλειμμα, διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Έχουμε φτάσει τώρα στην ε, Συμφωνία Πλαίσιο για την γονική άδεια. Θα σας παρακαλούσα οι συζητήσεις να γίνουν εκτός της αίθουσας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Συμφωνήσαμε σήμερα να έχουμε ανταλλαγή ε, απόψεων με τους ε, εμπειρογνώμονες. Ε, συμφωνήσαμε έτσι με την κυρία Μαρία Αρένα και καλωσορίζω τους εμπειρογνώμονες την κυρία Μαρία Τορζάριο Πάλμα, τον κύριο Καπρίτα, την κυρία Μίλσε και την κυρία Άντσε Κέρσταϊν. Δέκα λεπτά έχει στη διάθεσή της η καθηγήτρια Μαρία Τορζάριο Πάλμα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Πίσω μου κάθεστε, <laughs> αυτό δεν το συνηθίζουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία διαφάνεια, ελπίζω να εμφανιστεί. Δεν έχει εμφανιστεί. Θα έπρεπε να έχουν εμφανιστεί οι διαφανειές μου. Ζητώ συγγνώμη. Yes, I have. I should be there. So, wer macht, wer kümmert sich denn bitte um diese Präsentation? Ποιος ασχολείται με την τεχνολογία?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 Ωραία, θα προσπαθήσω να προχωρήσω χωρίς την ε, παρουσίαση και τις διαφάνειες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω μία έρευνα σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας 2010-18 και ο βασικός λόγος ύπαρξης της έρευνας αυτής αφορά η έκθεση για το συγκεκριμένο θέμα η οποία παρουσιάστηκε προετοιμάστηκε από τους ε, εμπειρογνώμονες για την ισότητα ε, των δύο φίλων και παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Ο βασικός, η βασική εστίαση του, της έρευνας αυτής έχει να κάνει με την εφαρμογή και έχουμε και κάποιες προτάσεις σε σχέση με ε, την εφαρμογή και μια, και μια ε, ε, καλύτερη ε, ενσωμάτωση της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας ε, στο μελλοντικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά. Θα περάσω κατευθείαν ε, στις εξελίξεις της έρευνας και της έκθεσης εφαρμογής. Όπως είπα, η έρευνα μου βασίστηκε σε μία έκθεση από το ε, δίκτυο ισότητας των φύλων ε, και η βάση είναι οι εθνικές εκθέσεις ε, τις οποίες υποβάλλουν οι διάφοροι εμπειρογνώμονες. Αν δούμε καταρχάς το εθνικό πλαίσιο της οδηγίας αυτής, της έκθεσης για την ισότητα των φύλων και την εφαρμογή της, Έχουμε μία καλή θεώρηση για τα ζητήματα της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως η εφαρμογή της οδηγίας 18 ε, του 2010 ε, λαμβάνει χώρα. Τρεις προκαταρτικές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, όλες οι χώρες έχουν πολύ περίπλοκα προγράμματα με σκοπό την προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας ε, και την πρόθεση... Α, εμφανίστηκαν και οι διαβάνειές μου. Έχω φτάσει ήδη σε αυτή τη σελίδα στο εθνικό ε, πλαίσιο. Όλες οι χώρες λοιπόν έχουν ε, πολύ περίπλοκα προγράμματα για ε, την ε, προώθηση της συμφιλίωσης οικογενειακής και της επαγγελματικής ε, ζωής και αυτό είναι ένας, μια εξήγηση για το λόγο για τον οποίο αυτή η οδηγία η 18 του 2010 δεν εφαρμόστηκε από πολλά κράτη-μέλη γιατί θεωρούν ήδη ότι η εθνική νομοθεσία είναι ήδη συμβατή με την ενωσιακή νομοθεσία. Συμπεριλαμβάνει λοιπόν αυτή η οδηγία συγκεκριμένε νέους διακανονισμούς ε, ε, εργασίας και ε, της μερικής απασχόλησης και μάλιστα σε μερικαία προγράμματα ο εντοπισμών συγκεκριμένων μέτρων ποικίλει από κράτος σε κράτος και επίσης αποκλίνει από την ενωσιακή προσέγγιση. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει ε, διαδοχικά ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ξεκινώντας από την άδεια Μητρότητα και μετά ε, με την ύπαρξη δικαιωμάτων συμφιλίου οικογενειακή και επαγγελματική ζωής, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε πάρα πολλά κρατημέλη. Αυτό το οποίο ισχύει σε σχέση με τη γονική άδεια και τις άλλες μορφές άδειας είναι ότι σε μερικές χώρες υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ ε, των ε, αδειών, αλλά σε άλλες χώρες ε, η γονική άδεια είναι μια περιεκτική μορφή άδεια η οποία μπορεί να συμπεριλάβει και την άδεια μητρότητας και σε μια τρίτη ομάδα χωρών η άδεια μητρότητας είναι η περιεκτική άδεια η οποία μπορεί να συμπεριλάβει τη γονική άδεια το συμπέρασμα από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις είναι ότι όχι μόνο το όνομα αλλά και το περιεχόμενο της γονικής άδειας σε εθνικό επίπεδο είναι συχνά πολύ διαφορετικό από την έννοια της γονικής άδειας ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ε, βλέποντας ε, τα θέματα που καλύπτει η γονική άδεια στο πλαίσιο της οδηγίας, ε, πώς τα κράτη-μέλη έχουν αντιμετωπίσει το θέμα και πώς έχουν ε, μεταγράψει στην ομοθεσία τους όλα αυτά τα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η γονική άδεια σε σχέση με άλλες άδειες που έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Σε μερικά κράτη-μέλη ισχύει το εξής. Η γονική άδεια πρέπει να ακολουθεί την άδεια μητρότητας και η διάρκεια της εξαρτάται από την διάρκεια της άδεια μητρότητας. Σε μερικά κρατημέλη υπάρχει επίσης ε, μία ξεχωριστή άδεια πατρότητας, αλλά σε άλλες χώρες η άδεια πατρότητας, αυτό που θα αποκαλούσαμε ε, ε, άδεια πατρότητας, είναι απλώς ένας χρόνος, μια άδεια από από την εργασία σε μερικές χώρες ε, ο όρος γονική άδεια είναι πολύ συγκεκριμένο, σε άλλες χώρες είναι ευρύτερος και συμπεριλαμβάνει και άλλου είδους ε, άδεια για φροντίδα του παιδιού. Ε, σε σχέση με το τι αποκαλείται γονική άδεια σε άλλες χώρες. Όσον αφορά τη διάρκεια της άδειας της γονικής, πολλά κράτη-μέλη χρειάστηκε να αλλάξουν την ομοθεσία τους για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με την ελάχιστη διάρκεια των τεσσάρων μηνών. Σε ε, πολλά ε, κράτη-μέλη η, γονική άδεια είναι ακόμη μεγαλύτερη, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τους τέσσερις μήνες. Η διάρκεια της γονικής άδεια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και κάτι το πολύ ενδιαφέρον είναι η σύγκριση της ε, μέγιστης επίσημης άδειας βάση νομοθεσίας και η πραγματική διάρκεια της γονικής άδειας. Όλοι οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν στα συμπεράσματά τους ότι η διάρκεια της άδειας έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την αποζημίωση. Σε μερικές χώρες η άδεια είναι αμοιβόμενη αν είναι αμοιβόμενη για μικρότερη διάρκεια από τη διάρκεια ε, που ε, προβλέπεται, ε, τελικά η άδεια που λαμβάνεται είναι μόνο αυτή που είναι με αμοιβή. Σε γενικές γραμμές η γονική άδεια είναι το δικαίωμα του κάθε γονέα. Όμως μερικοί γονείς έχουν μια γενική αρχή μεταφοράς, δυνατότητας μεταφοράς, ενώ σε άλλες χώρες ισχύει το αντίστροφο, δεν ισχύει η αρχή της δυνατότητας μεταφοράς και υπάρχει μία εξαίρεση, μία συγκεκριμένη άδεια, ε, ε, η οποία δεν μπορεί να ληφθεί ως άδεια γονική. Τώρα, ε, οι τρόποι εφαρμογή της γονικής άδεια είναι διαφορετικές, αλλά σε γενικέ ε, γραμμές ο κανόνας είναι μία ε, πλήρης γονική άδεια. Ένα, κάτι άλλο είναι ε, το θέμα ε, των διακρίσεων στις περισσότερες χώρες ε, ε, ε, προβλέπεται το δικαίωμα του να επανέλθει κανείς στην ίδια εργασία που είχε πριν με την ίδια αμοιβή. Αυτό που είναι διαφορετικό όμως είναι η ίδια η αμοιβή και αυτό είναι πραγματικά ένα βασικό ζήτημα. Η αμοιβή μερικές φορές ε, δεν δίδεται από τον εργοδότη αλλά από κάποιο επίδομα στα περισσότερα κράτη-μέλη. Όμως με πολύ διαφορετικούς όρους ε, το ποσό μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο ποσό ή ένα ποσοστό της ε, αμοιβή του μισθού του εργαζομένου. Αλλά μπορεί να ε, είναι ένα κατά ε, ποσό και σε μερικές χώρες δεν ε, πληρώνεται καν. Υπάρχουν και άλλα μέτρα στο πλαίσιο της γονικής άδειας σε μερικές χώρες, όπως για παράδειγμα ειδικό διακανονισμός του χρόνου εργασίας, υπάρχουν διάφορα μέτρα και υπάρχει και η άδεια πατρότητα. Σε μερικά κράτη-μέλη, λίγα, υπάρχει μια ξεχωριστή άδεια πατρότητας. Η άδεια για υιοθεσία επίσης υφίσταται, είτε ως ξεχωριστή άδεια, είτε ε, ως εφαρμογή απλώς των διατάξεων για την άδεια μητρότητας ε, ή για ε, την γονική άδεια στους γονείς τους θετούς. Η επιπλέον άδεια μπορεί να ισχύει ε, μόνο σε περιπτώσεις ε, ανωτέρας ε, βίας. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και για τη δική μου την έρευνα. Όσον αφορά την πρακτική χρήση της γονικής άδειας, οι διατάξεις αυτές, οι επίσημες ε, αφορούν το κατά πόσο λαμβάνεται η γονική άδεια ή όχι. η ορη είναι η εξή. Υπάρχει άλλη γονική άδεια που να έχει λάβει άλλο μέλος οικογένειας και δεύτερον κατά πόσο ε, το βάρος της άδεια είναι μοιρασμένο στου δύο όχι. Σε κάποια κρατημένη, ή όχι. Τα, σε κάποια κράτη-μέλη ε, η γονική άδεια παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Ε, όλοι οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η άδεια ε, η γονική συνήθως λαμβάνεται από την μητέρα και μάλιστα αναφέρονται και διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες ε, αναφέρουν επίσης ότι η εθνική νομοθεσία σε γενικές γραμμές ε, συμμορφώνεται με την ε, ενωσιακή νομοθεσία. Υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις, υπάρχει θετική προσέγγιση όσον αφορά την άδεια που λαμβάνουν οι πατέρες Υπάρχουν όμως δύο βασικές αδυναμίες που εντοπίζονται. Πρώτον, η σχέση μεταξύ των διαφόρων αδειών, η οποία δεν είναι καθόλου σαφή σε μερικές χώρες. Και δεύτερο πρόβλημα που θεωρείται και βασικό ζήτημα για την πρακτική χρήση της γονικής άδειας, είναι το θέμα της αμοιβή. Ένα ακόμη ε, λεπτό θα ήθελα ε, να χρησιμοποιήσω το χρόνο σας γιατί καθυστέρησα κιόλας να αρχίσω το δεύτερο σημείο της παρουσίασής μας, εντάχει, κάποιες, ενδείξεις, κάποιες υποδείξεις για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε ε, από εδώ και στο εξή. Η άδεια μητρότητας και η γονική άδεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα με διαφορετικές ε, πηγές ε, στην συνθήκη, η ασφάλεια και η υγεία και ε, κοινωνική προστασία, έχει να κάνει με τις γυναίκες ή με τις γυναίκες και τους άντρες και έχουν έναν διαφορετικό ε, κύριο στόχο. Η άδεια μητρότητας είναι το θέμα, ε, καλύπτει το θέμα της ασφάλειας και της υγείας των γυναικών στο χώρο εργασίας και η γονική άδεια έχει να κάνει με τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν δούμε αυτές τις δύο οδηγίες, ε, βλέπουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων υπάρχει ένα κοινό σημείο. Συνδέονται με την αρχή της ισότητας των φύλων. Η οδηγία για την άδεια μητρότητας δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια και την υγεία, αλλά έχει να κάνει και με την προστασία της ε, ισότητας των φύλων, δεδομένου ότι ε, θεωρείται άμεση διάκριση το να μην επιτρέπεται η άδεια μητρότητας. Από την άλλη, γονική άδεια αφορά όχι μόνο τη συμφιλίωση, αλλά και μία ισορροπία ε, στην ισότητα των φύλων ε, στο πλαίσιο της συμφιλίωσης. Οπότε λοιπόν η ισότητα των φύλων είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτών των δύο οδηγιών. Παρά το γεγονός λοιπόν ε, του ότι υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, αυτές οι δύο οδηγίες ε, ε, θέλουν να επιτύχουν το ίδιο στόχο, δηλαδή την συμφιλίωση οικογενειακού, οικογενειακού και επαγγελματικού βίου στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων. Η πρότασή μας θα ήταν συνεπώς να υπάρχει η αρχή της ισότητας των φύλων εντός των συνθήκων ως ε, ε, επίσημη βάση για ε, τη μελλοντική νομοθεσία και είναι διαφορετικό από αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό θα ήταν η δική μου πρόταση. Βεβαίως, μια τόσο διαφορετική προσέγγιση θα καθιστούσε το σύστημα πιο ε, ε, συνεπές, πιο διαφανές, θα ήταν πιο σαφής ο στόχος και θα υπήρχε μικρότερος κίνδυνος αντιπαραγωγικών μέτρων. Θα ήταν και ευκολότερο ε, να εφαρμοστεί και η ε, άδεια πατρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Χόρχε Καμπρίτα που κάθεται πίσω μου. Δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω μία παρουσίαση με διαφάνειες. Ελπίζω να μπορέσουμε να τη δούμε. Εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Εργασίας ε, στο Δουβλίνο και η παρουσίασή μου βασίζεται σε έρευνες ε, που κάναμε πρόσφατα σχετικά με την ε, γονική άδεια στην Ευρώπη καθώς και μία έκθεση σχετικά με τις προϋποθέσεις για την άδεια μητρότητας. θα... Αναφερθώ λοιπόν σε αυτές τις έρευνες αλλά και σε άλλες που επικεντρώνονται στη γονική άδεια. Η παρουσίασή μου ασχολείται κυρίως με πέντε ε, θέματα. Θα εξετάσουμε τους πιο σημαντικούς ορισμούς, θα κοιτάξουμε ε, τον χρόνο εργασίας ε, και την ισορροπία ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, τον ε, βαθμό στον οποίο ε, χρησιμοποιείται η γονική άδεια και κάποια άλλα διάφορα θέματα. Όσον αφορά λοιπόν ε, το πλαίσιο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο άρθρο 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρεται ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην ε, άδεια μητρότητας ε, και ε, την πληρωμένη άδεια μετά από την γέννηση παιδιού. Θα πρέπει να θυμόμαστε και την σχετική οδηγία του 1992 που από τη φύση της περιορίζεται στις γυναίκες. Σημαντικό είναι ε, να έχουμε κατά νου και τις κατευθυντήρες ε, γραμμές 2020 ε, που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της στρατηγικής 2020 όπου τονίζεται η εφαρμογή πολιτικών στην απασχόληση που να προωθούν την ίση μεταχείριση. Έχουμε επίσης την αναδιατύπωση οδηγίας του 2006 όπου καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να προωθήσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και τον ε, συνδυασμό επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Και κατόπιν έχουμε την ε, οδηγία του 2010 σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια της γονικής άδειας, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ε, δεν υπάρχει εδώ ελάχιστη αποζημίωση σχετικά με το εισόδημα που είχε κανείς πριν. Έχουμε ένα δίκτυο όπου ζητάμε από τους ε, ανθρώπους στα κράτη-μέλη να μας δώσουν ε, στοιχεία. Δεν υπάρχουν εναρμονισμένα δεδομένα. Από τα λίγα δεδομένα που υπάρχουν, διαπιστώνουμε ότι το χαμηλό ποσοστό εκμετάλλευσης ε, της γονικής άδειας από τους πατέρες είναι γενικό. Υπάρχει μια αύξηση, αλλά πολύ αργή. Γίνεται δηλαδή όλο και περισσότερη χρήση της ε, άδειας πατρότητας, αλλά παρόλα αυτά πολύ λίγοι χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή. Ορισμοί. Είναι σημαντικό εδώ να θυμηθούμε τα τρία είδη άδεια. στην άδεια μητρότητας, που ε, είναι ε, πάυση εργασίας για τη μητέρα πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι ε, ένα διάστημα σωματικής ανάρρωσης. Κατόπιν έχουμε την γονική άδεια που γενικά θεωρείται δικαίωμα των εργαζομένων που είναι μια δυνατότητα που δίνεται και στους δύο γονείς για να φροντίσουν το παιδί μετά τη γέννα του παιδιού και συνήθως ακολουθεί το διάστημα της άδεια μητρότητας και κατόπιν έχουμε την άδεια πατρότητας που είναι μια σύντομη άδεια μόνο για τον πατέρα μετά τη γέννηση παιδιού που του επιτρέπει ε, να ε, περάσει ε, το χρόνο του με το παιδί και τη σύζυγο. Να σας δείξω κάποιες διαφάνειες που βασίζονται στην έρευνα, την ευρωπαϊκή έρευνα των συνθήκων εργασίας. δείχνει τον χρόνο που δαπανούν τα δύο φύλλα ανά εβδομάδα σε διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι η μη πληρωμένη εργασία κυρίως ε, πραγματοποιείται από γυναίκες, ενώ οι άνδρες ε, έχουν περισσότερη πληρωμένη εργασία. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ε, φροντίδα μικρών παιδιών ή άλλων ενηλίκων, αυτό γίνεται κυρίως από τις γυναίκες και θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Όσον αφορά τους ε, άγαμους ε, γονείς, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ε, την υποστήριξη ενός συντρόφου και έτσι η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εδώ βλέπετε ακριβώς το ίδιο, τον χρόνο ε, πληρωμένης και απλήρωτης εργασίας ανά εβδομάδα. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι γυναίκες που έχουν μερική εργασία εργάζονται σχεδόν τον ίδιο χρόνο με τους άντρες ε, που έχουν θέση πλήρους απασχόλησης, αν λάβουμε υπόψη τον ε, χρόνο μετακίνησης και τον χρόνο απλήρωτης εργασίας. αυτά τα στοιχεία είναι του 2015, βλέπουμε μια μικρή αλλαγή, αλλά οι μεγάλες διαφορές παραμένουν. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι άνδρες ασχέτως της ηλικίας τους αναφέρουν ε, χειρότερο τέριασμα ανάμεσα στις επαγγελματικές ε, και ιδιωτικές δραστηριότητες. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί οι άνδρες το ισχυρίζονται αυτό. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι γυναίκες οργανώνουν την ε, επαγγελματική τους ζωή γύρω από τον ιδιωτικό τους βίο, ενώ οι άνδρες επικεντρώνονται κυρίως στον επαγγελματικό βίο. Αυτό ίσως εξηγεί τη διαφορά εδώ. Αν κοιτάξουμε λοιπόν ε, το τι άδειε ε, υπάρχουν σε διάφορες χώρες, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σα σε μια σειρά χωρών όπου υπάρχουν ε, κάπως ειδικέ συνθήκες. Έχουμε την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Μάλτα, όπου δεν υπάρχει άδεια πατρότητας, υπάρχει γονική άδεια, αλλά απλήρωτη άνευ αποδοχών. Και έχουμε εδώ άλλες τέσσερις χώρες, ε, Ελλάδα, κάτω χώρες, ε, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η γονική άδεια είναι άναφα αποδοχών και η ε, άδεια πατρότητας δεν είναι υποχρεωτική. Και θέλω να σας δείξω τον αντίκτυπο που, που έχει η δομή των αδειών στην οικογενειακή ζωή. Στις χώρες αυτές ε, βλέπουμε ότι το σύστημα φαίνεται να μην προωθεί τον ρόλο του πατέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπε σήμερα το πρωί, αναφέρθηκε στον ρόλο του πατέρα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, τίθενται κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα. Κάποια από τα πιο βασικά ευρήματα που θα ήθελα να ε, μοιραστώ μαζί σας είναι το ποσοστό χρήσης της άδεια πατρότητας. Με βάση λοιπόν τις έρευνες που ανέφερα για την άδεια πατρότητας, μητρότητας και την γονική άδεια, βλέπουμε ότι η εθνική νομοθεσία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό χρήσης της άδειας. Η προλαλή σα το ανέφερε αυτό. Ο τρόπος όπου είναι οργανωμένη η γονική άδεια παίζει σημαντικό ρόλο. Και επίσης σημαντικό ρόλο παίζει το ρόλο το αν οι διατάξεις είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Πολύ σημαντική είναι η οικονομική υποστήριξη. Οι χώρες που ε, δίνουν μεγαλύτερο ποσοστό αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της άδεια ε, έχουν και αυξημένη χρήση. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, διότι χρειάζονται περισσότερη στήριξη για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις άδειε αυτές, διότι αλλιώς δεν θα χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος. Υπάρχουν κάποιες στρατηγικές για να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην χρήση γονικής άδειας και άδειας πατρότητας. Κάποιοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή διότι φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή ότι δεν θα ξαναβρούν την ίδια δουλειά όταν επιστρέψουν. Εμείς ως ε, διεύλος επικοινωνίας ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζομένους θέλουμε να διασφαλίσουμε κατά τη διάρκεια της άδειας ε, να επικοινωνεί ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, κάτι που δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας. Επίσης, ε, σε επίπεδο χώρου εργασίας, η ευελιξία και οι πρακτικές των εργοδοτών ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σημασία δηλαδή έχει όχι μόνο η νομοθεσία, αλλά και το πώς εφαρμόζεται στον χώρο εργασίας. Αυτό επηρεάζει το πώς γίνονται αντιληπτές ε, αυτές οι άδειε. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι σαφείς, θα πρέπει να είναι ευέλικτοι οι κανόνες, θα πρέπει να είναι απλοί ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητοί από τους πιθανούς χρήστες. Θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με την ε, διαθεσιμότητα ε, υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και οι πολιτικέ ισορροπίες ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην ευελιξία κυρίω απέναντι στι γυναίκε, αλλά ε, δεν τονίζεται επαρκώ η ενθάρρυνση των ανδρών. Και οι δραστηριότητε στον τομέα τη ισότητας των δύο φύλων ε, θεωρούνται μάλλον ε, επιμορφωτικές και σε λιγότερο βαθμό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αλλάζουν την πραγματικότητα. Νομίζω ότι ήδη έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Θα κλείσω με τα εξής. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Είδαμε ότι υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά την κατανομή χρόνου εργασίας για την απλήρωτη ε, και την πληρωμένη εργασία ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Ε, οι άντρε ε, θεωρούν ότι είναι δύσκολο να συνδυάσει το επαγγελματικό και οικογενειακό βίο. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, κίνητρα κατά τη διάρκεια τη άδεια, ε, διότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση για το αν θα χρησιμοποιήσει κανείς τη δυνατότητα αυτή ή όχι. Σημαντικό είναι να συζητώνται τα πράγματα αυτά στον χώρο εργασίας διότι εκεί εφαρμόζεται ο νόμος και εκεί μπορεί να προκύψουν οι δυσκολίες. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι παράγοντες κλειδιά στη διαδικασία αυτή, είτε στη διαμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής, αλλά και στην εφαρμογή στον χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε διοικητικό και οικονομικούς περιορισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους πατέρες να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα της γονικής άδεια και θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές που να αλλάζουν την πραγματικότητα και όχι ε, να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε ενημερωτικές πολιτικές. Εδώ βλέπετε τα εξώφυλλα ε, δύο εντύπων που δημοσιεύθηκαν φέτος. Υπάρχουν ακόμα κάποια αντίτυπα έξω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τους επιστημονικούς μας συνεργάτες από το EPRS και το Aerofan για την πολύ σημαντική πληροφόρηση που μας έδωσαν και βεβαίως όλα αυτά είναι καλό να γίνονται εντός του χρόνου. Λοιπόν, έχουμε τώρα τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των συνδικάτων. Η κυρία Μίλτς από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων, η TUC, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τηρήσω το χρόνο μου, γιατί πολλά θέματα έχουν ήδη καλυφθεί. Ο συνδυασμός εργασίας και οικογενειακής ζωής δεν είναι καινούριο εδώ και δύο δεκαετίες ε, περίπου, δηλαδή από τότε που είχαμε την ε, οδηγία για την γονική άδεια, ασχολούμεθα με το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε τι προκλήσεις έχουμε, κατά πόσο λαμβάνεται αυτή η γονική άδεια, κατά πόσον εγγυόμεθα σε ενωσιακό επίπεδο αυτό το συνδυασμό εργασίας και οικογενειακού βίου, αλλά και πώς τώρα βγαίνοντας από την κρίση θα έχουμε ένα συνεκτικό νομοθετικό πλέγμα για να εφαρμοστεί η δυνατότητα αυτή. Νομίζω ότι η εφαρμογή της οδηγίας είναι επιτυχία και καταδεικνύει τη σημασία του ενωσιακού κοινωνικού διαλόγου. Η συμφωνία αυτή αναθεωρήθηκε δύο φορές και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει χαμηλό ποσοστό λήψης, αυτό μας ανησυχεί. Πιστούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σφαιρικό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο. Το νέο ε, συγγνώμη, ο νέος οδικός χάρτης για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στο συνδυασμό εργασίας οικογένειας είναι σημαντικός για να διαμορφώσουμε ουσιώδη δικαιώματα που θα εξασφαλίσουν τη λήψη αυτής της άδειας. Το βασικό θέμα είναι που θα μας οδηγήσει αυτός ο δικός χάρτης για το συνδυασμό εργασίας-οικογένειας. Θα διατηρήσει το status quo ή θα το βελτιώσει. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Όλες οι μελέτες, όλη η έρευνα έχουν καταδείξει ότι το βασικό θέμα για την αύξηση της λήψης της άδεια είναι η αμοιβή της. Από την οπτική μας γωνία η αμοιβή είναι το βασικό σημείο, η βασική προτεραιότητα. Σε ορισμένες χώρες ξέρουμε ότι δίνεται ένα καταποκοπήν ποσό. Αυστρία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Σλοβακία, Σουηδία και άλλες χώρες. Σε άλλα κράτη-μέλη οι παροχές αυτές πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ποσοστό του μισθού. 30% στην Ιταλία, 60% στην Πολωνία, 67% στη Γερμανία, 70% στη Φιλανδία, 80% στην Αυστρία και 100% στη Δανία και την Πορτογαλία αλλά για μικρότερη περίοδο. Σε σχεδόν όλες τις άλλες χώρες δεν υπάρχει αμοιβή Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα Ιρλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Η γονική άδεια είναι άνευ αποδοχών. Και στις περισσότερες περιπτώσεις όπου είναι αμοιβόμενοι, είναι δημόσια δαπάνη μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και όχι οι εργοδότες. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ακόμη πιο σημαντικό Μερικά από τα τελευταία στοιχεία που έχουμε λένε ότι η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών κοστίζει 325 δις, δηλαδή γύρω στο 2,5% του ΑΕΠ της Ένωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι γυναίκες δεν ε, καταφέρνουν να εργαστούν όπως θα έπρεπε, κοστίζει αυτό 30% του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει λοιπόν να το δούμε το θέμα αυτό. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να λαμβάνουν και οι άνδρες γονική άδεια όπως και οι γυναίκες. Οι ε, γονείς λοιπόν είτε είναι βιολογικό το τέκνο είτε θετό θα πρέπει να μπορούν και οι δύο να λαμβάνουν την άδεια. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι μόνο μικρή είναι η αύξηση της λήψης από τους άνδρες. Από 3% στο 4% μεταξύ του 2005 και του 2013. Άρα το ποσοστό λήψη από τους άνδρες είναι πολύ χαμηλό. Καταλήγοντας. Κυρίως ανησυχούμε για το ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει ένα ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο πλήρες που να βασίζεται στην αμοιβή της γονικής άδειας και σε μια ενιαία προσέγγιση που να συνδυάζει όλες τις διάφορες άδειες μητρική, πατρική, για θετά παιδιά και την άδεια για αυτούς που φροντίζουν για άλλους. Μια νέα προσέγγιση λοιπόν που να καλύπτει όλα τα είδη τέτοιας άδειας σε όλες τις φάσεις της απασχόλησης ενός εργαζόμενου. Είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη γενιά σάντουιτς. Δηλαδή τα άτομα που χρειάζεται να ασχοληθούν και με τα παιδιά τους και με ηλικιωμένα άτομα που έχουν ανάγκη φροντίδας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η Άντια Γκέρνσταϊν από το Business Europe. Και εκείνη πέντε λεπτά. Ευχαριστώ εκπροσωπώ την οργάνωση Business Europe. Και προέρχομαι από τη Γερμανική Συνομοσπονδία Εργοδοτών και Επιχειρήσεων, BDA. Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας, διαπιστώσαμε ότι συνολικά η εφαρμογή της και η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο είναι ικανοποιητική. Με βάση αυτά που μας λένε οι οργανώσεις μέλη μας στις περισσότερες χώρες, η οδηγία αυτή θεωρείται ότι έχει μεταγραφεί, έχει μεταφερθεί με ικανοποιητικό τρόπο, με ομαλό τρόπο. Οι οργανώσεις μας δεν μας ανέφεραν ε, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην πορεία μεταφοράς. Η εθνική κοινωνική εταίρου δεν συμμετείχαν αυτόματα. Έχει να κάνει με την κατάσταση στις χώρες μέλη, στα κράτη-μέλη αλλά σε ορισμένε περιπτώσεις υπήρξαν είτε επίσημες είτε ανεπίσημες διαβουλεύσει. Και ο τρόπος συμμετοχή τους έχει να κάνει με τις ε, διαδικασίες τριμερούς διαβούλευση που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη για διάφορα θέματα, για ευρύτερα θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με γονική άδεια και φροντίδα για τα παιδιά. Αυτό δείχνει ότι συνεχίζεται ο διάλογο με τι κυβερνήσει για διάφορα είδη άδεια Αυτό το ακούσαμε και σε μια προηγούμενη ομιλία. Και για όλους τους διακανονισμούς που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μεταφορά της οδηγίας σχετίζεται με πολλά θέματα που συζητώνται τώρα σε διάφορες ε, χώρες για το συνδυασμό εργασίας οικογένειας και η λήψη της άδειας σχετίζεται πολύ στενά με την αμοιβή που ε, ποικίλει πολύ από χώρα σε χώρα. Αλλά από ό,τι μάθαμε εμεί δεν είναι ο μόνο παράγμα που επηρεάζει τη λήψη. Ο τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, οι πατέρε ζητούν περισσότερη ευελιξία για τι ώρε εργασία. Και η δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων δυνατοτήτων βοήθεια στην φροντίδα για τα παιδιά παίζει επίσης μεγάλο ρόλο. Αυτά μας λένε οι οργανώσεις μέλη μας. Τώρα πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε αυτή τη συγκυρία δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να προβλεφθούν νέες μορφές άδειας σε ενωσιακό επίπεδο. Όπως νομίζω ότι προέκυψε και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις Πρέπει να γίνουν βαθιές αλλαγές ε, στην κοινωνία μας. Και στη Γερμανία από όπου προέρχομαι έχουμε ακόμη αυτό τον όρο Gartenmutter. Τι σημαίνει αυτό. Τις ε, γυναίκες που θέλουν να κάνουν και παιδιά και να κάνουν καριέρα. Όσο υπάρχουν τέτοιοι όροι δεν βελτιώνει την κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης, μία νέα σχέση μεταξύ μητέρα και, μητέρας και πατέρα. Αυτό δεν θα το επιτύχουμε με νομοθετήματα. Πρέπει να αλλάξει επίσης η συμπεριφορά στους χώρους εργασίας. Και οι δύο γονείς θα πρέπει να απαιτούν νέες μορφές εργασίας που να τους επιτρέπουν ακριβώς να συνδυάσουν την εργασία με την ε, φροντίδα των παιδιών. Αυτό θα γίνει εκεί συγκεκριμένα, στους χώρους εργασίας. Δεν μπορεί να επιτευχθεί με νομοθετήματα. Και αυτό διαπιστώνουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά όχι επαρκώς. Κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν καλή βρεφονιμφιακή σταθμή και άλλες δυνατότητες φροντίδας. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι απλώς πάρκινγκ. Πρέπει να είναι χώροι όπου να τους δίδεται εκπαίδευση υψηλού επίπεδου για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, προσαρμοσμένοι τις ανάγκες τους. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι στα διάφορα κράτη-μέλη έχει πολύ διαφορετικές μορφές η γονική άδεια, άρα δεν είναι πλήρως συγκρίσιμη η κατάσταση. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη είναι ο συσχετισμός των διαφόρων αδειών. Σχεδόν όλες οι χώρες έχουν αναπτύξει πολύ περίπλοκα, συστήματα για να προστατεύσουν τις εγγύους και τη μητρότητα και για να προωθήσουν τον συνδυασμό εργασίας οικογένειας. Αυτά τα συστήματα έχουν να κάνουν βέβαια με τα δικαιώματα και τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης κάθε κράτους μέλους και το επίπεδο προστασίας εργασίας, τις σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων, την ε, προσαρμοστικότητα των ωραρίων εργασίας κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τους εμπειρογνώμονες Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την Μαρία Αρένα, για πέντε λεπτά, αλλά αν τα καταφέρετε σε τρία λεπτά, ακόμα καλύτερα. Merci, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις σας. θα ήθελα να κάνω καταρχάς μία διαπίστωση που θα μας βρει όλους σύμφωνους, είτε είμαστε πολιτικοί ηθήνοντας, είτε είμαστε επιστήμονες, είτε είμαστε κοινωνικοί εταίροι, είναι ότι σήμερα ζούμε τη μεγαλύτερη διάκριση στην Ευρώπη, δηλαδή μία διάκριση που πλήττει και τους άνδρες και τις γυναίκες. Δηλαδή σήμερα οι άνδρες πατέρες οι που επιθυμούν να γίνουν πατέρες ε, είναι θύματα διάκρισης γιατί δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα με τις γυναίκες, δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακού και ε, επαγγελματικού βίου. Μας το είπαν και οι εμπειρογνώμονες άλλωστε. Υπάρχει μια αίσθηση μεταξύ των ανδρών σήμερα στην Ευρώπη ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ισότητα μεταξύ του ιδιωτικού και του επαγγελματικού βίου. Επομένως, αγαπητοί κύριοι, θα εργαστούμε υπέρ ε, στο πλαίσιο το, της, γονικής, γονικής άδειας. Δεύτερη διάκριση κατά των γυναικών. Πιστεύετε ότι κάτω επιλογή οι γυναίκες αποφασίζουν ε, το, ε, ε, επιλέγουν να κάνουν το μεγαλύτερο τμήμα ε, μία αμοιβόμενη εργασία ε, από εσά, πιστεύετε ότι είμαστε πιο μισάνθρωποι από εσά. Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Επομένω, αυτό είναι μία διάκριση και η διάκριση αυτή μα ακολουθεί σε ολόκληρη τη ζωή μα, ε, γιατί υπάρχει διάκριση στο χώρο εργασία, στο πλαίσιο τη σταδιοδρομία. Δείτε τι καριέρε των γυναικών στους μισθούς αλλά και στη σύνταξη. Ε, επειδή χρειάστηκε να κάνουμε λοιπόν τις επιλογές μας από την αρχή, από τη στιγμή που αποφασίζουμε να γίνουμε μητέρες, εκτός εάν θα ήθελε ε, το ποσοστό γεννήσεων της η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ακόμη χαμηλότερο και δεν νομίζω ότι αυτό είναι στόχος κανενός, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε αυτή την πορεία διάκρισης και υπάρχει ένα φαινόμενο σήμερα στην Ευρώπη 100% διάκριση, δηλαδή 100% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι θύμα διακριτικής μεταχείρισης και επομένω είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα τι μπορούμε να κάνουμε για να μην συμβαίνει αυτό. Γιατί γιατί και από απόψεως οικονομικής και από απόψεως κοινωνικής αυτή η διάκριση στοιχίζει, στοιχίζει, γιατί όταν δεν είναι κανεί ε, ικανοποιημένο από τη ζωή του, έχει αντίκτυπο στην υγεία του. Σήμερα οι στατιστικέ ε, τη κατάθλιψη, ε, γι' αυτό υπάρχουν, υπάρχει μια συναισθηματική υγεία πολύ αλλοιωμένη σήμερα στην Ευρώπη. Υπάρχουν επίση όμω και οικονομικέ συνέπειε. Όλε οι μελέτε μα δείχνουν ότι αν υπήρχαν περισσότερε γυναίκε στην αγορά εργασία και λιγότερη διάκριση εναντίον του, θα είχαμε περισσότερε μεγαλύτερο ΑΕΠ. Μεγαλύτερο ΑΕΠ. Εντάξει, δεν θα μπορώ να τα συνδέσω και άμεσα, αλλά μερικές φορές είναι το μόνο επιχείρημα που πιάνει τόπο. Ε, μιλάμε σήμερα ε, για ε, συμφωνίες όπως η ε, TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μιλάμε για αύξηση 0,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αν υποθέσουμε ότι θα συμβεί αυτό. Το να έχουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας θα ε, επέτρεπε αύξηση του ΑΕΠ της τάξεως του 3%. Μια άλλη επιστημονική ανάλυση την οποία μπορούμε να αμφισβητήσουμε. Αλλά όταν βλέπουμε σήμερα ε, την πίεση που υπάρχει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτήν την TTIP ε, πραγματικά μου κάνει εντύπωση όταν βλέπουμε λοιπόν την έλλειψη δημιουργικότητας ε, που επιδεικνύουμε όσον αφορά τις γυναίκες και τη συμμετοχή τους στην ε, αγορά εργασίας και βλέπουμε πόση δημιουργικότητα επιδεικνύουμε σε επιχειρηματικό επίπεδο ε, λέμε ότι όχι, ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει νομοθεσία, ότι ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει βελτίωση. Μου κάνει ε, εντύπωση το να λένε οι εργοδότες ότι δεν θέλουν να υπάρξει 3% αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οπότε εγώ ζητώ και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω όλα στην έκθεσή μου, Ζητώ λοιπόν να υπάρχει μία ε, συνεκτική ε, προσέγγιση σε σχέση με το θέμα της μητρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας. Ζητούμε να υπάρξει μία ρήτρα αναθεώρησης ε, της γονικής άδειας. Το θέμα της αμοιβή επίσης είναι σημαντικό γιατί είδαμε ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και στο ποσοστό απορρόφησης αλλά και σε σχέση με τα φύλλα. Δηλαδή όσο το ε, θέμα τίθεται σε οικονομικούς όρους ε, οι γυναίκες είναι αυτές που παίρνουν περισσότερο άδειε μητρότητας. Ε, το θέμα της γονικής άδειας, της διάρκειάς της είναι σημαντικό. Τέσσερις μήνες είναι επαρκής, μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα της παιδικής ηλικία που δεν τελειώνει ίσως στα 8 χρόνια, ότι η παιδική ηλικία υπερβαίνει τα 8 χρόνια. Το θέμα της νομοθεσίας και της άδειας πατρότητας, εμείς ζητούμε ε, το θέμα αυτό να αποτελεί ένα εργαλείο ε, και νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε ότι όταν υπήρχε η άδεια πατρότητα στα κράτη-μέλη και λαμβανόταν, ε, τότε οι άντρες όλο και περισσότερο λάμβαναν άδεια πατρότητας. Συμφωνώ με την Business Europe σε σχέση με αυτό που είπε τα συνοδευτικά μέτρα των παιδικών σταθμών της φροντίδας των παιδιών παιδιών ε, της φύλαξης των παιδιών. Είναι γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνεπώς αυτά τα συνοδευτικά μέτρα και για παιδιά που ασθενούν ε, και για ε, παιδιά ε, ε, πριν από το σχολείο, δηλαδή σε επίπεδο παιδικών σταθμών, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό και έχει άμεση σχέση με τους δείκτες ισότητας στο χώρο εργασίας. Πρέπει να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια εξελικτική πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδού λοιπόν τα έξι σημεία τα οποία θα ήθελα να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου για το καλό όλων των γυναικών, των ανδρών, αλλά και των επιχειρήσεων και της Ευρώπης ευρύτερα. Ευχαριστώ. Maria σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές, ένα λεπτό ο καθένας, ο Κρίστοφ Χέκμαν είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τονίσουμε το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα μας επιτρέψει να συνδυάσουμε καλύτερα τον ιδιωτικό με τον επαγγελματικό βίο. και που θα διευρύνει τα δικαιώματα της πατρότητας. Δεν είναι μόνο κάτι το οποίο επιθυμούν οι πολίτες, αποτελεί και δική μας προτεραιότητα. Νομίζω ότι σημαντική καινοτομία της οδηγίας του 2010 ήταν η ε, αύξηση της γονικής άδειας, της άδειας πατρότητας από τρεις σε τέσσερις μήνες. Που δεν μπορεί, ο τέταρτος μήνας δεν μπορεί να μεταβαστεί στην ε, σύζυγο. Έτσι ενθαρρύνουμε τους άντρες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην οικογενειακή ζωή. Σήμερα όμως ακούσαμε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις ώστε να ενθαρρύνουμε τους άνδρες να χρησιμοποιούν την άδεια πατρότητας. Σημαντικές είναι επίσης οι περιπτώσεις ανθρώπων που ε, εργάζονται με μερική απασχόληση ή μέσω γραφείων που παρέχουν υπηρεσίες. Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά στο θέμα της γονικής άδεια. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να εξετάσουμε τις διαφορές που υπάρχουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και επίσης χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτή την πολύ σημαντική έκθεση και θα συνεργαστώ στενά με την κυρία Αρένα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Κέρι και για ένα λεπτό επίσης. Ακούσαμε πολλά για την αδιαμητρότητα, την αδιαπατρότητα, τη γονική άδεια. Γίνονται σημαντικά βήματα εδώ. Και αυτό που δεν ισχύει καθόλου στον όρο αυτό είναι ότι πρόκειται για άδεια, είναι δουλειά. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν στα κράτη-μέλη πρέπει να πληρώσουν οι γονείς για τη φροντίδα των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς ε, κλπ, ε, τότε θα πρέπει να μιλάμε για δουλειά. Δεν είναι άδεια, δεν είναι διακοπές η γονική άδεια. Και θα έπρεπε να συζητάμε το τι θα έπρεπε να πληρώνεται αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη όμως. Γι' αυτό σας καλώ να γίνει μια σημαντική τροποποίηση σε όλες τις εκθέσεις ε, που συζητάμε. Να μην μιλάμε για parental leave, να μιλάμε για δουλειά των γονέων, όχι για άδεια. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Χάρκιν. Είναι στούπερ. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu queria, em primeiro lugar, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε. Συχνά Μπερδευόμαστε και εμείς όταν μιλάμε για την ε, οδηγία για την άδεια μητρότητα ε, και την οδηγία για τη γονική άδεια. Σημαντικό είναι να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά. Και θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση. Όταν μιλάμε για ευελιξία στην εργασία, όταν μιλάμε για την γονική άδεια και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την επιστροφή των γονέων στον χώρο εργασίας, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ε, για τι πράγμα μιλάμε. Υπάρχει ο δικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την νέα οδηγία και αναφέρεται η ευελιξία ως λύση. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει στην ε, μη εγγύηση κάποιων σημαντικών δικαιωμάτων. Γιατί, διότι η ευελιξία θα πρέπει να θεωρηθεί δικαίωμα των γονέων. Δεν θα πρέπει να χάνουν ε, δικαιώματα κοινωνικά, εργασιακά, ε, όσον αφορά την αμοιβή κλπ. Δεν θα πρέπει δηλαδή οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την ευελιξία ως δικαιολογία. Σημαντικό ερώτημα εδώ είναι το θέμα των χρημάτων που λαμβάνει κανείς, διότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της οδηγίας. Το να είναι κανείς γονέας είναι κοινωνική ευθύνη και θα πρέπει να προστατεύεται ε, η, ιδιότητα αυτή. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Μόνικα Βάνα. Δεν είναι εδώ η Μόνικα Βάνα. Τότε η Λάουρα Ατζέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε αυτή την ε, δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις διαφόρων ε, φορέων που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ επίσης τη Άλφα Μαρία Αρένα ε, με την οποία φυσικά προσβλέπουμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης αυτής της έκθεσης. Έχω ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις και θέματα που θα ήθελα να τονίσω. και ε, προτάσεις ε, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Πάνω απ' όλα, η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων για όλες τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε κατηγορηματικά. Αυτό θα επιτρέψει επίσης ε, να αυξηθεί και η γεννητικότητα. Να βοηθήσουμε λοιπόν τα δικαιώματα και των ανδρών και θα βοηθήσουμε έτσι την επιστροφή στην εργασία και των ανδρών και των γυναικών μετά την γονική άδεια. Και σε αυτό θέλω να επιμείνω. Υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα του κειμένου. Για παράδειγμα, η επέκταση της γονικής άδειας εάν ε, ε, επιτρέψουμε όπως γίνεται σε ορισμένες χώρες να επεκταθεί μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανατροφή των παιδιών, για την εκπαίδευσή τους, για να ασχοληθούν οι γονείς με τα παιδιά. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά παράλληλα είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί αν δεν υπάρξουν επαρκείς οικονομικές ε, ενισχύσεις, μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, επαρκής ε, βοήθεια επαρκής αμοιβή για να ενισχύσουμε αυτή τη δυνατότητα λήψης ε, μεγάλου διαστήματος γονικής άδεια και να προτείνουμε και πολύ συγκεκριμένα μια ισότιμη κατανομή των βαρών που αφορούν την φροντίδα ανατροφή των παιδιών δηλαδή και οι δύο γονείς να ασχολούνται στο μέτρο του δυνατού ισότιμα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εργασία το να κανείς Νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο αγαθό, κάτι που μας έχει δοθεί. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους γονείς στις επιλογές τους, να τους επιτρέψουμε να γίνουν καλοί γονείς. Γιατί ξέρετε ότι στην Ήπειρό μας ε, πολλές οικογένειες ε, παρετούνται του δικαιώματος να ε, αναθρέψουν παιδιά, να αποκτήσουν παιδιά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Γιατί λοιπόν να μην προβλέψουμε ένα εγγυημένο οικογενειακό εισόδημα για ε, τα πρώτα έτη της ζωής των παιδιών ανεξάρτητα από την απασχόληση. Να έχουμε δηλαδή κάποιες μορφές κοινωνικής προστασίας για αυτές τις καταστάσεις. Για παράδειγμα μέσω ενός οικογενειακού εισοδήματος μπορούμε να το παρουσιάσουμε με διαφορετικούς τρόπους αυτό να το δούμε. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να επιτρέψουμε τους γονείς, στους γονείς να παίξουν το ρόλο τους ως γονείς πρέπει να τους δώσουμε τις προϋποθέσεις. Και βεβαίω θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφό μα για τι πρώτε ενδείξει που μα έδωσε. Πρόεδρο. Ντομινίκ Μαρτνά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα σε εκπλήξω, αλλά είμαι πολύ πιο φιλόδοξος ε, από τη Μαρία Αγενά και συμφωνώ περισσότερο με την προηγούμενη ακριβώς ομιλήτρια. Προφανώ άδεια μητρότητα για τη γυναίκα που έχει γεννήσει κάποιε εβδομάδε πριν, 6 με 8 εβδομάδε μετά. Μία γονική άδεια για τη μητέρα ή τον πατέρα που να μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 2 ή 3 έτη ηλικία του παιδιού, μέχρι να μπει στο σύστημα σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης. Και κάτι ακόμη. Επειδή συμφωνώ με τη συνάδελφο του EFDD, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα οικογενειακό μισθό, οικογενειακό γονικό μισθό για τη μητέρα ή τον πατέρα μέχρι να φτάσει σε, στην ενηλικίωση το τελευταίο τους παιδί. Δεν συμφωνώ καθόλου με την κυρία Ρένα και πολλούς άλλους. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι υπάρχουν άνδρες ή γυναίκες που θα προτιμούσαν να αναθρέψουν το παιδί τους μέχρι να ενηλικιωθεί παρά να πηγαίνουν να δουλεύουν για ένα άθλιο μισθό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ωραία. Η Ντανούτα Γιαζολέτσκα. Εντάξει, εντάξει, άλλοι δύο θα πάρουν το λόγο, αλλά μετά θα πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε τρία τέταρτα καθυστέρηση. Η Ντανούτα. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, γιατί έχει πολλές φορές ε, αναφερθεί ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση ή υποκατάσταση των μισθών ε, για όλους όσους παίρνουν αυτού του είδους τις άδειες μητρότητας, γονική, πατρότητας, ε, Υπάρχουν καλές πρακτικές ε, με ένα μείγμα ε, διαφόρων μέτρων. Μήπως θα μπορούσατε αυτό ε, να μας το πείτε. Τελευταία ομιλήτρια. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη θα ήθελα να τονίσω και να εστιάσω στο γεγονός ότι η περίοδος μητρότητας δεν είναι ακριβώς μία αμοιβούμενη χρονική περίοδος, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μία οικονομική υποστήριξη της μητέρας ή του πατέρα κατά τη διάρκεια της άδειας. Επαφίεται στο κράτος μέλος ποιο είναι το επίπεδο που θα αποφασιστεί και πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα στους γονείς με επιπλέον ε, υποστήριξη οικονομική για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Αλλά αν συγκρίνει κανείς τα κράτη-μέλη και τις συνθήκες που υπάρχουν, πρέπει να λάβετε υπόψη και το ποιότητα, την ποιότητα και την προσβασιμότητα άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η ποιότητα και η προσβασιμότητα των ε, ε, υπηρεσιών της υγείας ε, και των παιδικών σταθμών, είτε είναι δωρεάν είτε είναι με πληρωμή και ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών στις δύο περιπτώσεις. Διαφορετικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ο συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασιστεί σε κοινά ελάχιστα, σε κοινές ελάχιστες προδιαγραφές. Δεν είναι, διαφορετικό, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα μονολυθικό σύστημα. Ευχαριστώ για την ερώτηση της, για, της Ντανούτα. Θα παρακαλούσα τους ε, επιστήμονες που έκαναν τις παρουσιάσεις να ενημερώσουν την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Η έκθεση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, οπότε η Μαρία θα πρέπει να εργαστεί και κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών και στις 16 Μαρτίου θα εγκριθεί στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονές μας και τους εκπροσώπους του ETUC και του, της οργάνωσης Business Europe. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο το 6 που θα πρέπει να το συζητήσουμε 27 λεπτά οι στόχοι κατά της φτώχειας ε, λόγω των αυξανωμένων εξόδων για τα νοικοκυριά ο εισηγητής μας είναι ο Ταμάς Μέζοριτς ελπίζω να είναι σύντομος και οι εξίσου παρακαλώ Τάμας, πού είσαι, α εκεί ευχαριστώ πολύ σας παρακαλώ προς λέει ησυχία. Θα είμαι να τον ε, πιο σύντομος μπορώ, αλλά να σας εξηγήσω γιατί είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Η αρχική μας διαπίστωση που ελπίζω να την συμμεριζόμεθα πολύ εδώ είναι ότι η Ευρώπη αργά αλλά σταθερά δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους του 2020. Οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τουλάχιστον τους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας θα ωφελούσε την Ένωση και όλους, τους, όλους τις τους πολίτες. Ένα στοιχείο κλειδί, ίσως όχι το σπουδότερο, είναι τα έξοδα των νοικοκυριών. Όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο στοιχείο του κόστους για τα περισσότερα νοικοκυριά και για το μέσο νοικοκυριό είναι το κόστος της ενέργειας, τα καύσιμα. Το θέμα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προώθηση των ανανεωσίμων. Αυτός είναι νομίζουμε ένας απτός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για να στοχεύσουμε περισσότερο τη βοήθεια προς τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν έντονη ενεργειακή φτώχεια. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι είναι ένα ειδικό είδος φτώχειας αυτό, όπου υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Ο λόγος για τον οποίο πολλά φτωχά νοικοκυριά ξοδεύουν τόσα πολλά για καύσιμα ή γενικότερα για ενέργεια είναι επειδή το σύστημα θέρμανσής τους δεν είναι καθόλου αποδοτικό. Είναι παλιά και δαπανηρά συστήματα θέρμανσης. Αλλά η αντικατάστασή τους είναι ακριβή. Δεν μπορεί λοιπόν να την πληρώσει ένα φτωχό νοικοκυριό. Άρα ακόμη και αν αυξηθεί λίγο το εισόδημα ενός τέτοιου νοικοκυριού δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Γι' αυτό πιστεύουμε Χρειάζεται μια πιο συνολική προσέγγιση. Δηλαδή στοχευμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και στοχευμένα μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα βοηθούσε δηλαδή ο συνδυασμός αυτών των δύο. Ποιες είναι οι βασικές συστάσεις. Πρώτη, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη παράλληλα να εγκρίνουν αυτά τα ενοποιημένα πλαίσια καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας. Αυτό χρειάζεται γιατί είναι διαφορετικές αρμοδιότητες των δύο αυτών ε, φορέων. Και ακόμη στο εσωτερικό της Επιτροπής χρειάζεται εναρμόνιση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και των μέτρων αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης καλούμε τα κράτη-μέλη να προσυπογράψουν ένα μορατόριο για τη διακοπή παροχής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι καιρός να υπάρξει αυτό. Υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη. Αλλά κάποια κράτη-μέλη όπου οι κοινωνικές παροχές είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένες έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει σε όλα τα κράτη-μέλη. Καλούμε την Επιτροπή στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα να παρουσιάσει μια οδηγία πλαίσιο για το κατάλληλο ελάχιστο εισόδημα. Και τέλος χωρών τα κρατή-μέλη να διασφαλίσουν πιο αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ευρωπαϊκών περιφερειακών και επενδυτικών πόρων και από τι τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχέ, για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Πώ τώρα θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα μέσα. Δεν το αναφέρει το σχέδιο έκθεση όχι επειδή δεν έχουμε ιδέες για το πώς θα κινητοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, αλλά για τους κανόνες ε, που περιορίζουν το μήκος των εκθέσεων. Θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες με πιο συγκεκριμένες συστάσεις. Αλλά επίσης θα θέλαμε τις ιδέες των σκιωδών στην Επιτροπή μας και βεβαίως να τις συμπεριλάβουμε στην τελική έκθεση. Είμαι ανοιχτό για κάθε διαπραγματεύσει για οποιοδήποτε τμήμα του κειμένου. Νομίζω πως θα είναι φορά η συζήτησή μα. Τέλος. Το κείμενο αυτό οφείλεται και στην Καταλήν Τζίβα και τον Φίλιν Σούλτσε αλλά εάν υπάρχουν κάποιες ε, ανεπάρκειες ή ασάφειες εγώ αποκλειστικά είμαι υπεύθυνος αλλά μέσω αυτή τη ανταλλαγή απόψεων που θα κάνουμε τώρα πιστεύω ότι θα τις υπερβούμε. Ευχαριστώ και προσβλέπω και στη συζήτηση με του Κιώδη. Ευχαριστώ πολύ. ναι. Ευχαριστώ πολύ να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας σε επίπεδο έκθεσης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Εγώ θα κάνω μερικές παρατηρήσεις για την ώρα, τρεις παρατηρήσεις γενικής φύσεως. Δικαίως ε, η σημασία που αποδίδεται στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας ε, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο αυτό. Παρόλα αυτά, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχετε και περιορισμό όσον αφορά το ε, Μέγεθο του κειμένου. Υπάρχουν όμως στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης ε, και ε, της κοινωνικής στέγασης, της πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για τις φτωχέ οικογένειες με μεγάλη αύξηση των δαπανών τους για ιατρικέ υπηρεσίε. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά προβληματικό όπως επίσης και η πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες και αναφέρομαι για παράδειγμα στην κινητικότητα. Στις περιοχές της Υπέδρου η πρόσβαση ε, στην άδεια οδήγησης είναι μεγάλο πρόβλημα και συνεπώς είναι μεγάλο εμπόδιο για την έβρεση εργασίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κάτι ακόμη το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το αναφέρουμε περισσότερο είναι το ε, θέμα των παιδιών ε, στις οικογένειες, στις ε, φτωχές. Είναι σημαντικό να καθορίσουμε ορισμένες έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση όσον αφορά το ίσο ελάχιστο εισόδημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε γιατί διαφορετικά ε, θα συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα και τελικά θα δούμε ότι μιλάμε ε, με όρους μαύρου και άσπρου και ε, δεν θα μιλάμε καθόλου για το ίδιο πράγμα. Κάτι ακόμη, ένα στοιχείο ευρύτερη στρατηγικής είναι να προσπαθήσουμε από τη μία να είναι όσο το δυνατόν πιο συνενετικό το κείμενο γιατί έτσι θα είναι και πιο ισχυρό δεδομένου του προβληματισμού που υπάρχει αλλά και ένα κείμενο το οποίο θα μας επιτρέψει το συντομότερο δυνατόν να φτάσουμε στην εφαρμογή των πρακτικών και των αποφάσεων σε το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πολύ χαρά λοιπόν θα απαντήσω στην προσφορά σας για θετική συνεισφορά σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα στην Ήτρε, ψηφίζαμε επί σχεδόν δύο ώρες. Ε, φοβάμαι ότι δεν έχουμε διερμηνία προς τα φιλανδικά, θα ήταν ωραία να είχαμε. Στην ε, γραμματεία μιλώ, δεν με προσέχει όμως. Όταν είμαι σκιώδη συσυγήτρια θέλω πολύ να έχω φιλανδική διερμηνία διότι είναι πολύ πιο εύκολο να μιλώ στη μητρική μου. Θα προσπαθήσω όμως να τα πω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλό να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια. Και να φροντίσουμε για κοινωνική ένταξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας να έχει ασφαλή στέγαση. Η ενέργεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ από τη Φιλανδία έρχομαι, είναι σχετικά πλούσια χώρα. Εάν λοιπόν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως υπάρχει αναντιστοιχεία, αυξάνονται συνεχώς οι τιμές. Έτσι λοιπόν στα κέντρα των πόλεων είναι πολύ διαφορετικές οι τιμές από ό,τι αλλού. Ο σωστός σχεδιασμός λοιπόν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, κάτι που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες, σε πολλά μέρη της Ευρώπης, ήταν η φούσκα στις τιμές ε, ακινήτων και πολλές οικογένειες έχασαν το σπίτι τους και άλλοι πληρώνουν, πλήρωναν υπερβολικά μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους για να πληρώσουν το δάνειο, τελικά έχασαν το σπίτι τους και πάλι δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Αυτή λοιπόν η μεγάλη εξάρτηση από τα χρέη είναι μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι τράπεζες να κάνουν κάτι γι' αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να ασχοληθούν με το πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς δάνειο και να αγοράσει δικό του σπίτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που είναι χαμηλά τα επιτόκια. Τώρα είναι εύκολο να πάρει κανείς δάνειο. Αν αλλάξουν τα πράγματα όμως ή αν σκάσει η φούσκα, ε, τότε μπορεί να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα. Πάντως ε, θα πρέπει να είναι πιο ισχυρή η κοινωνική διάσταση και στις συστάσεις αναχώρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τους παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους στη φτώχεια. Όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο, αυτό είναι το θέμα, όχι μόνο το εισόδημα. Το θέμα είναι δηλαδή είναι αν έχει κανείς στέγη ή τα σε για τις μεταφορές, για το πόσιμο νερό ή για τη θέρμανση το χειμώνα. Νομίζω ότι μπορούμε να υπογραμμίσουμε κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου ε, οι γυναίκες ε, που ζουν πολύ καιρό με χαμηλές συντάξεις ε, όταν είναι χείρες, οι ηλικιωμένοι, οι φοιτητές, συχνά είναι δύσκολο να βρουν στέγαση οι φοιτητές, και μειονότητες ε, επίσης ε, στην ε, Φιλανδία. Τα νοικοκυριά με έναν γονέα είναι επίσης ομάδα κινδύνου και τώρα μάλλον θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους μετανάστες και την ανάγκη για κάποιο είδους στέγαση για όλους τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και που δεν ξέρουμε αν θα μείνουν για λίγο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. όσον αφορά το θέμα της ενέργειας σε σχέση με την φτώχεια. Θα σχολιάσω αργότερα πιο συγκεκριμένα, διότι μελετώ την κατάσταση σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Σε κάποιες χώρες είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το θέμα. Σε άλλες χώρες ε, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Εξαρτάται και από τα κοινωνικά επιδόματα. Πρόεδρος, ε, Έχουμε στη διάθεσή μας ε, μόνο 16 γλώσσες. Ε, το Κοινοβούλιο δεν μας ε, δίνει περισσότερες. Θα καλούσα λοιπόν την πολιτική σας ομάδα να θέσει το θέμα στο Προεδρείο. Ο Αρνεγκέρικε. Δύο λεπτά αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ω σκιώδης εισηγητή ε, τη πολιτική μου ομάδα, ε, Βρίσκω πολύ σημαντική την πρόταση αυτή, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί περιλαμβάνουμε εδώ την ε, πράσινη προσέγγιση στην ενέργεια σε μια έκθεση για την φτώχεια. Δεν άκουσα ούτε μία φορά τη λέξη οικογένεια. Είναι οι πρώτοι που επηρεάζονται από την φτώχεια λόγω έλλειψης τροφίμων, η ε, έλλειψης θέρμανσης, η ε, έλλειψης στέγασης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο θέματα και θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω μέχρι ε, να το καταλάβει το Κοινοβούλιο. Η εργασία των γονέων, η φτώχεια των γονέων και η φτώχεια των παιδιών ε, συνδέονται στενά μεταξύ τους ε, και θα πρέπει να είναι σαφές ότι μια οικογένεια με παιδιά κινδυνεύει κατεξοχήν από την φτώχεια. η δουλειά των γονέων ε, δεν πληρώνεται, δεν υπάρχει ελάχιστη αμοιβή, δεν πληρώνονται όπως πληρώνονται ε, οι βρεφονιπιακοί σταθμοί κλπ. Και ε, το κόστος ενός παιδιού είναι πολύ υψηλό. Ακόμα και αν δεν συμπεριλάβουμε τις δαπάνες για, την, για τις σπουδές. Θα θέλουμε να μιλάμε για μια κοινωνία αλληλεγγύης και η ανατροφή των γονέων είναι μια υπηρεσία προς ε, το κράτος. Φυσικά αγαπούν οι γονείς τα παιδιά τους, φυσικά είναι συναισθηματικό το θέμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αυτή, διότι ε, αλλιώς ε, θα χρεοκοπήσουμε κοινωνικά. Επίσης, η γραφειοκρατία ε, και μάλιστα αυτή που συνδέεται με τις Βρυξέλλες, με την Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη ε, δυσκολεύονται να, να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την ε, γραφειοκρατία. Και ο Έντμουν Στόιμπερ που υποτίθεται ότι θα ασχολιόταν με τη μείωση της γραφειοκρατίας δεν έχει καταφέρει να την μειώσει για τα νοικοκυριά μας. Θέλω 50% λιγότερη γραφειοκρατία για τα νοικοκυριά μας. Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να πω ότι ο μόνος που δεν εξήγησε τον χρόνο ομιλίας του σήμερα ήταν ο Ντέιβιτ Κάζα και εγώ έχω απελπιστεί. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Σε δύο λεπτά λίγα μπορεί να πει κανείς. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο σύντροφός μου ρολά. άρα δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά επιμένω ότι το θέμα αυτό αφορά τη φτώχεια λόγω των εξόδων των οικοκυριών. Δεν είναι μία μελέτη ενεργειακή πολιτική, ούτε για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν ξέρω αν ε, είναι ο στόχος κάποιον, αλλά όταν μιλάμε για τους ε, που, για αυτούς που πραγματικά υποφέρουν από φτώχεια, ο τρόπος που μιλάμε είναι λιγάκι εξευτελιστικός. Πρόκειται για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ηλεκτρικό και προσπαθούν παράνομα να πάρουν. Ορισμένοι δεν έχουν ούτε καν σπίτι. Πρέπει να καταλάβουμε πώς έχει η κοινωνική πραγματικότητα στην οποία εργαζόμεθα. Η κατάσταση επίσης είναι Πώ αντιμετωπίζουμε βράχη πρόθεσμα. Ένα θέμα είναι ενεργειακή πολιτική που έχει να κάνει με την ε, ενεργειακή ανεξαρτησία κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με τον εισηγητή μας που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ως βάση. Γιατί κοιτάξτε, ορισμένα τα υποστηρίζω. Είμαι στην διαπολιτική ομάδα για την φτώχεια και καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη φτώχεια. Δεν υπάρχει φτώχεια για τα μωρά και τους μεγάλους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά τη φτώχεια μόνο μέσω ενός οικογενειακού εισοδήματος. Μετά θα έχουμε καλύτερη κοινωνία, καλύτερη ενέργεια κτλ. Αλλά γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε για ένα ελάχιστο εισόδημα που φυσικά θα προσαρμόζεται στο επίπεδο κάθε χώρας και κάθε κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν και τα υπόλοιπα θα τα πω μέσω τροπολογιών, αρκούμε στο να πω ότι θα πρέπει να αγωνιστεί για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Καταπολέμησης της Φτώχειας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ένα σπίτι το σώστε όποιος έχει σπίτι που είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό ή το οποίο μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συνδυάζονται. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καλύτερο τρόπο καταπολέμηση φτώχεια είναι ένα οικογενειακό εισόδημα. Λίν Πάουλεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα δύο λεπτά. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας, για αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δικαίως αναφέρεται το γεγονός ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω όσον αφορά το, τη φτώχεια και δεν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2020. Γνωρίζω ότι στην Ιρλανδία η ε, πολιτικές λιτότητας ε, έχουν διπλασιαστεί από το 2008 και συμφωνώ με το θέμα του ενεργειακού κόστους και ε, των οικοκυριών αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι σκιώδεις συζητητές. Θα ήθελα λίγο περισσότερες αναφορές στο κόστος του νερού. Ξέρουμε ότι είναι όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με 6% των ε, εσόδων των οικοκυριών ε, που πηγαίνει στο νερό, οπότε θα ήθελα να αναφέρετε και αυτό. Και κάτι ακόμη για να συμφωνήσω με την ποιότητα και την παροχή κοινωνική στέγαση στην Ιρλανδία, επειδή γνωρίζω, έχουμε 15.000 παιδιά που ζουν σε τέτοιου είδους στέγαση προσωρινά, κάτι το οποίο σημαίνει κόστος που οδηγεί σε περαιτέρω φτώχεια και όσον αφορά τις πολιτικές ε, λιτότητας ε, οι οποίες προωθούνται σε χώρες ε, που βρίσκονται σε προγράμματα όπως η Ιρλανδία, θα υπάρξει ένα, υπάρχει, υπάρχει ένα έγγραφο βασικό για το οποίο εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η Λόρα Ατζέα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την προσέγγιση του επί του θέματος αυτού που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, θα ήθελα να ε, προβάλλω κάποιες αντιρρήσεις εγώ δεν βλέπω κανένα, καμία σύνδεση με το θέμα της απασχόλησης και των κοινωνικών προβλημάτων. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο ενεργειακό ζήτημα. Οπότε Αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι που δεν έχουν ένα σπίτι, γιατί το μεγαλύτερο τμήμα των ε, φτωχών οικογενειών δεν έχουν καν ε, μία εστία το ενεργειακό πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα στάδιο μετά από το βασικό τους πρόβλημα. Θα έπρεπε λοιπόν να ασχοληθούμε πρώτα με το πρώτο πρόβλημα. Προφανώς θα συμμετέχω στην εργασία αυτή. Θα ήθελα να αναφερθούμε στη μη κατάσχεση της πρώτης ε, κατοικίας, ειδικότερα στις ε, ε, περιπτώσεις χωρών που έχουν πολλά προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να χάνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι και ε, ε, δεν μπορούν να πληρώσουν το, το νίκη τους. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των ε, βραχυπρόθεσμων μέτρων και του κατεπήγοντος που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα επιγόντως τώρα. Θα υποβάλω τροπολογίες, ελπίζω να τις αποδεχθεί ο εισηγητής. Το σχολείο, ε, η παιδική σταθμή δεν πρέπει να πληρώνουν οι οικογένειες ε, οι οποίες ε, δεν μπορούν καν δημόσιες, δημόσιους παιδικούς σταθμούς να πληρώσουν. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των οικογενειών και των, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Γιατί άμα, δείτε κανείς, τα, άμα δει κανείς τα αριθμητικά στοιχεία, είναι τρομακτική η κατάσταση. Στις χώρες όπου υπάρχει κρίση, οι πρώτες δαπάνες ε, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά είναι ιατρικές, η ιατρική φροντίδα πολλές οικογένειες δεν μπορούν καν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Ε, δεν μπορούν να έχουν ιατρική περίθαλψη για τα παιδιά τους. Δεν είναι δυνατόν ε, να μην υπάρχουν βασικές υπηρεσίες για τις οικογένειες της φτωχές αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της φτώχειας. Νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Συμφωνώ με τους λογαριασμούς ε, του ηλεκτρικού, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Δεν είναι εδώ ο Μπιτσότο. Ωραία. Οπότε κλείνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Προθεσμίες. 17 Νοεμβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή στις 17 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα. Το 7 δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε. Ο εισηγητής είναι εδώ. Θα μπορούσαμε να αναβάλουμε το θέμα αυτό για το απόγευμα μετά τις ψηφοφορίες. Αλλά δεν θα είναι παρόν ο εισηγητής. και τρεις κοιόδης ε, εισηγητές ε, δεν θα είναι παρόντες το απόγευμα. Οπότε συμφωνώ με τον εισηγητή Ερίκε Καλβέτ Τσαμπον ότι η συζήτηση θα γίνει με τους κοιόδης εκτός συνεδρίας Επιτροπής διότι έτσι μπορούν να συζητήσουν και περισσότερο σε βάθος. Συμφωνείτε με αυτή τη διαδικαστική πρόταση για να αποφύγουμε αυτό το σκόπελο. Ναι. Τόμας. Ένα λεπτό. Αν μιλήσει ο καθένας μας είναι τρεις ε, Λοιπόν τέσσερις. Έχουμε τέσσερις ε, παρόντες. Θα μπορούσαμε τέσσερα λεπτά. Ναι. Δεν σε πιστεύω όμως λέει ο πρόεδρος. Δεν πιστεύω. Ενρίκε. Ένα λεπτό. Και μετά οι άλλοι επίση σύντομα. Όχι, δεν είναι δυνατόν με ένα λεπτό. Δεν θα ήταν σωστό. Αλλά βεβαίως, βεβαίως, να ασχοληθούμε σε συναντρίαση των ε, σκιωδών. Δεν θα ήταν διανοητικά έντιμο να το συζητήσουμε σε τρία λεπτά. Μα αυτό θεώρησα κι εγώ. Έτσι ξέρω ότι λειτουργεί ο Ενρίκε. Οπότε σας παρακαλώ να το κάνουμε έτσι. Να το συζητήσουν οι σκιώδεις οπότε θα μπορέσει να είναι και ο Ενρίκε και θα μπορέσει να μιλήσει όπως πρέπει για να εξηγήσει το θέμα. Αυτό θα έχει επαρκή χρόνο. Συμφωνούμε? Ωραία. Οπότε διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Λοιπόν, για την έκθεση του Ενρίκε 17 Νοεμβρίου 12 η ώρα για τροπολογίες ε, η προθεσμία και στις 11 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Και άλλους λοιπόν πρέπει να δουλέψει στις διακοπές. Λοιπόν θα τα ξαναπούμε στις 3.